So, Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Ξαναρχίζουμε και συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας και με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω την Προεδρεύουσα του Συμβουλίου για θέματα υγείας, την κυρία Τρινιδάδ Χιμένες. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πολιτική υγείας είναι σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας. Και η Ισπανική Προεδρία για τους επόμενους έξι μήνες έχει ένα πρόγραμμα για αυτό το τομέα και έχουμε και εμείς πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Πολλές εκθέσεις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 για να μου δώσετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις γενικές γραμμές του προγράμματος της Ισπανικής Προεδρίας σε θέματα υγείας. Πρόκειται για τιμή και ικανοποίηση μεταξύ άλλων, γιατί η Ισπανία είναι μια χώρα η οποία είναι διαφυσβήτηκτα ευρωπαϊκά, είναι υπέρ του ευρωπαϊκού οράματος και είναι δεσμευμένη ε, για το σχέδιο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος από αυτή την οπτική γωνία αναλαμβάνουμε λοιπόν το έργο της Προεδρίας με ευθύνη και με ενθουσιασμό. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, διότι με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης Λισαβόνας ανοίγεται ένας νέος, ε, μια νέα περίοδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα όμως είμαστε καθόλου αδιατεθειμένοι και σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να ε, οδηγήσουμε σε αίσιο σε ένα πρόγραμμα εργασίας το οποίο είναι πολύ ε, φιλόδοξο και το οποίο έχουμε προετοιμάσει από κοινού με το Βέλγιο και την Ουγγαρία βάσει του νέου συστήματος των τριών προεδριών ε, βάσει των αρχών της αλληλεγγύης, της ευθύνης και της συνεργασίας. Κυρίες και κύριοι, η Ισπανική Προεδρία θέλει να συνεχίσει να εργάζεται για μια Ευρώπη ισχυρή, ενωμένη, πιο αποτελεσματική, πιο ολοκληρωμένη, πιο αλληλέγγυα και ταυτόχρονα πιο εύπορη. Σε θέματα υγείας αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να στοχεύσουμε στις αρχές και τις ε, αξίες που είναι κοινέ και που συμμεριζόμαστε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε όλα τα συστήματα υγείας να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού και κυρίως στις ανάγκες των ασθενών. Αυτές οι κοινέ αξίες και αρχές οι οποίες έχουν καθοριστεί στη ε, δήλωση του Συμβουλίου του ε, Ιουνίου του 2006 θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο των εργασιών μας στη διάρκεια της Προεδρίας. Δηλαδή, θέλουμε να επισημάνουμε όλα όσα ε, θεωρούμε ως την προμετωπίδα του μοντέλου της υγείας στην Ευρώπη, δηλαδή ε, την ισότητα, την αλληλεγγύη και την πρόσβαση σε, μια, ε, σε υπηρεσίες υγείας ασφαλής και καλής ποιότητας. Όλα στα πλαίσια ενός οικοδομήματος, ε, ενός χώρου υγείας, ο οποίος θα είναι κοινός για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πεπισμένοι ότι πρόκειται για στοιχεία τα οποία είναι ιδιαίτερω χρήσιμα για την αρμονική ανάπτυξη και την συνεκτική ανάπτυξη των διαφορετικών συστημάτων υγείας των κρατών μελών. Επιπλέον θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάποιες αλλαγές οι οποίες αλλάζουν την κοινωνία μας ε, με πολύ ουσιαστικό τρόπο στις τελευταίες δεκαετίες. Καταρχάς αναφέρομαι στις δημογραφικές αλλαγές. Μιλάμε για μια ευρωπαϊκή κοινωνία που έχει και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, ε, που γυράσκει ταχύτατα, αυξάνοντας ταυτόχρονα και την... Ε, ε την κυριαρχία των χρόνιων ασθενειών. Επίσης αναφέρομαι και στις συνεχείς τεχνολογικές ε, προόδους που μας ε, επιτρέπουν να βελτιώσουμε την έρευνα και την ε, ποιότητα της υγείας όποτε χρειαστεί. Γι' αυτό ακριβώς επιμένω ότι έχουμε ετοιμάσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στη σημασία των κοινωνικών παραγόντων της υγείας, στην όθηση για το e-health και την ε, δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων μεταξύ άλλων. Επιπλέον, θα ήθελα επίσης να επαναλάβω ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας δεσμεύεται να εργαστεί για να έχουμε συνένεση μεταξύ όλων των κρατών μελών για την οδηγία για τις ε, διομαθοριακές υπηρεσίες υγείας. Γι' αυτό και στις επόμενες μέρες έχω προβλέψει να ε, συζητήσω με τον νέο Επίτροπο, να μάθω την άποψή του για το θέμα και από εκεί και πέρα, από πλευράς Προεδρίας, να εργαστούμε για να προχωρήσει αυτό το ζήτημα. Κυρίες και κύριοι, θεωρούμε ότι η κοινοτομία στη δημόσια υγεία η επαγρύπνηση των ε, διαφόρων κοινωνικών παραγόντων για την υγεία και η εξαφάνιση, η εξάλληψη των ανισοτήτων θα πρέπει να αποτελεί βασικό στρατηγικό σημείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό το σκοπό θα αφιερώσουμε το άτυπο ε, συνέδριο Υπουργών Υγείας που θα γίνει στη Μαδρίτη στις 22 και 23 Απριλίου σε θέματα καινοτομία στη δημόσια υγεία και θα γίνει και μία διάσκεψη προπαρασκευαστική εμπειρογνωμόνων. Επίσης, έχουμε ε, συγκαλέσει και μία υπουργική διάσκεψη για την πρόθεση του e-health στη Βαρκελόνη στις 15 ε, από τις 15 έως τις 18 Μαρτίου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής αποτελούν στοιχείο κλειδί για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την καινοτομία, την ποιότητα και τη συνοχή των ε, ε, συστημάτων υγείας μας. Και είμαι βέβαιη ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όλοι στο γεγονός ότι το e-health είναι ένα στρατηγικός άξονας τον οποίο θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς θα χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε τις επενδύσεις και κυρίως να δώσουμε τη δυνατότητα για μια διαχείριση ποιότητας. Αν όμω έπρεπε να σταθώ σε μια πολύ συγκεκριμένη πτυχή του προγράμματο τη Ισπανική Προεδρία σε θέματα αν οποία οδηγία θα έλεγα ότι ο κοινό μα στόχο είναι να έχουμε μια νέα οδηγία, ευρωπαϊκή οδηγία ποιότητα και ασφάλεια σε θέματα δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων η οποία οδηγία θα περιλαμβάνει όχι μόνο τα κοινά στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα ταυτόχρονα και όλες τις καλύτερες ε, πρακτικές ε, τόσο οργανωτικές όσο και από πλευρά συνδρομής από τα διάφορα κράτη-μέλη τα οποία έχουμε συγκεντρώσει τόσα χρόνια που ασχολούμαστε στον τομέα, με τον τομέα αυτό της ιατρικής. Η Ισπανία θέλει να προσφέρει την πείρα της γιατί διαθέτει ένα πολύ οργανωμένο μοντέλο δωρεάς και μεταμεσχεύσεω οργάνων το οποίο βασίζεται σε αυτές τις αξίες και τις αρχές που σας ανέφερα στην αρχή της παρέμβασής μου. Δηλαδή, η αλληλεγγύη, η συνοχή, η ποιότητα και η καινοτομία αλληλεγγύη και ισότητα, διότι κανένας πολίτης δεν θα μπορέσει να αποτελέσει αντικείμενο διάκρισης για μεταμόσχευση, για λόγους κοινωνικής προέλευσης ή ε, τόπου διαμονής. Συνοχής, γιατί πρόκειται για ένα συντονισμένο σύστημα από τα κεντρικά και στο οποίο συμμετέχουν μέσα από ένα καινείο σύστημα όλες οι περιοχές της χώρας μας. Ποιότητα γιατί το μοντέλο ε, προσφέρει κάθε χρόνο παραμέτρους αριστείας σε κάθε έναν από τους δείκτες λειτουργίας του. Και καινοτομία γιατί καταφέραμε να ενσωματώσουμε όλες τις επιστημονικές προόδους που έχουν γίνει στον τομέα αυτό με επιτυχία και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις όπως είναι για παράδειγμα η ε, μεταμόσχευση ε, προσώπου ή ε, η δωρεά μεταξύ ζώντων. Ε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το μοντέλο ε, έχει αποδείξει ότι είναι μεγάλο ενδιαφέροντος και θα γίνει και κάποια επίσκεψη στην Ισπανία πριν από την διάσκεψη που θα κάνουμε στη Μαδρίτη της 23 Μαρτίου και είμαι βέβαιη ότι θα μπορέσουμε μεταξύ μας να τεθεί πολύ γρήγορα σε ισχύ αυτή η οδηγία την οποία ε, επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή, τη συζητάμε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα όσοι έχουν γίνει και γίνονται επί του θέματος. Η Ισπανική Προεδρία θα εργαστεί ε, προκειμένου να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και συνένεση για το θέμα αυτό και οι αξίες που σας ανέφερα πριν να παραμείνουν ε, στην οδηγία. Κυρίες και κύριοι, πέρα από τα στρατηγικά θέματα θα ήθελα να αναφέρω επίσης και κάποια άλλα στοιχεία του προγράμματος της Προεδρίας τα οποία θα σταθούμε με πιο εντατικό τρόπο. Καταρχάς, στον τομέα των φαρμάκων. Η Ισπανική Προεδρία θα συνεχίσει τις εργασίες που έκαναν οι προηγούμενες προεδρίας, η Τσεχική και η Σουηδική, αναθεώρησης του νομοθετικού πακέτου για τα φάρμακα, κυρίως τις ε, οδηγίες και τους κανονισμούς για τα παραποιημένα φάρμακα και την φαρμακοεπαγρύπνηση. Και ε, στόχος μας είναι να έχουμε μια πιθανή συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2010. Οι άτυπες συναντήσεις με τους εισηγητές ε, των αντίστοιχων εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ιδιαίτερως ικανοποιητικές και είμαι βέβαιη ότι θα καταφέρουμε να έχουμε κείμενα τα οποία θα είναι κατάλληλα για να ενισχύσουμε το βασικό μας στόχο που είναι η ασφάλεια των φαρμάκων. Δεύτερον, στον τομέα της διατροφικής ασφάλειας, η Ισπανική Προεδρία θα εστιάσει κυρίως στη συνέχεια της ανάπτυξης του νομοθετικού προγράμματος, κυρίως ε, σε θέματα ενημέρωσης κατανοητών και νέων τροφίμων, βάσει και των εργασιών που ήδη έχει κάνει η Σουηδική Προεδρία. Επίσης θα θέλαμε να δώσουμε μια σημαντική όθεση στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για προβλήματα που σχετίζονται με τη διατροφή, ε, την παχυσαρκία, ε, το να είναι κάποιος υπέρβαρος και όλα αυτά περιλαμβάνονται στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2007. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και λαμβάνοντας υπόψη και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για δράσεις για, να, για την πρόληψη των ε, καρδιακών παθήσεων, θα εργαστούμε στα πλαίσια του Συμβουλίου για μία πρόταση για τη μείωση της κατανάλωσης ε, άλατος και της υγείας. Και τρίτον, θα θέλαμε να δώσουμε ε, μια νέα όθηση στην ε, κλινική αριστεία και στην ε, συνέχεια της παροχής υγείας, κυρίως στον τομέα των χρόνιων ασθενειών που τις μη μεταδιδόμενες, οι οποίες είναι μεγάλη συχνότητα, όπως για παράδειγμα οι καρδιακές παθήσεις ή η ψυχική υγεία. Στόχος μας είναι να είναι κοινέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι βέλτιστες πρακτικές περιλαμβάνοντας κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές υπηρεσίες για τα ε, άτομα τα οποία πάσχουν από τις ασθένειες αυτές και τις οικογένειές τους βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα της ε, ε, θεραπείας ε, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, έχουμε διασφαλίσει, έχουμε οργανώσει διάφορα πράγματα, για να, διάφορες δράσεις για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ασφάλειας των ασθενών, ε, κυρίως ε, το θέμα της, των ασθενειών που σχετίζονται με την ιατρική περίθαλψη και την αντιμικροβιακή αντοχή και την καταπολέμηση φυσικά του AIDS. Κυρίε και κύριοι, όπω σα είπα και στην αρχή, θα αντιμετωπίσουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει διάφορε δραστηριότητε και διάφορε συνεδράσει. Είναι φιλόδοξο γιατί θέλουμε να έχουμε μια Ευρώπη η οποία θα είναι προετοιμασμένη και θα έχουμε ω βασικέ αξίε την ισότητα και την ευημερία και τις δυνατότητες για όλους τους πολίτες. Γι' αυτό ακριβώς ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ε, συμμεριστούμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία που μας προσφέρει η νέα συνθήκη της Λισαβόνας, την οποία ξεκινάμε τώρα. Να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι πιο αποτελεσματική, αλλά κυρίως και μια Ένωση που θα είναι πιο σχετική με τους πολίτες. Αυτό είναι ο βασικός μας τελευταίος στόχος και είμαι βέβαιη ότι εσείς που αντιπροσωπεύετε τη φωνή των σχεδόν 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αυτοί είναι αυτοί που θα πρέπει να αποτελούν το βασικό άξονα για όλες μας τις δράσεις. Μπορείτε φυσικά ε, να βασιστείτε σε μένα. Είμαι καθόλου διατεθειμένη να συνδιαλλαγούμε παντού και ανα πάσα στιγμή και στις χώρες μας και εδώ και δεσμεύομαι να είμαι πιστή στα θεσμικά όργανα. Αυτό ε, με υποχρεώνει να κάνω η θέση μου ως Προεδρεύουσα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και τώρα είμαι στη διάθεσή σας, ε, κύριε Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Πρώτη φορά έρχεστε στην Επιτροπή μας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείχνετε τη δέσμευση της Ισπανικής Προεδρίας. Έχετε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ε, χαίρομαι ε, γιατί έμεινε στο πρόγραμμα εργασιών σας το θέμα της διασυνοριακής ε, φροντίδας, γιατί είναι πολλά τα εκατομμύρια των πολιτών στην Ευρώπη που διαμένουν σε μεθοριακές περιοχές και ενδιαφέρονται και έχουν πολλές ελπίδες για αυτή τη νομοθεσία. Μεγάλος ο κατάλογος των ομιλητών και ξεκινώ με τους συντονιστές. Τρία λεπτά παρακαλώ. Πέτερ Λίζε είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Καλώ ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε εδώ τα λέω ισπανικά, αλλά τα υπόλοιπα θα σα τα πω γερμανικά. Για τις μεταμοσχεύσεις έχω να πω ε, κάποια σημεία κύριε Υπουργέ. Είναι πολύ θετικό το ότι το έχει συμπεριλάβει η Ισπανία. Είναι πρωτοπόρος η Ισπανία όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στις μεταμοσχεύσεις οργάνων. Και από την εμπειρία σας μπορούμε να διδαχθούμε κι εμείς. Δύο συγκεκριμένα σημεία. Στο άρθρο 18 ε, γίνονται διάφορε συζητήσει και ξέρετε ότι προτείνεται μια τροπολογία γιατί θέλουμε όλοι να είμαστε εξίσου καλοί με την Ισπανία. Αλλά όπω και στο ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να αντιγράφουμε το στυλ των άλλων. Σε άλλες χώρες υπάρχουν κάποιες δομές οργανωμένες ε, που θέλουμε να τις βελτιώσουμε αλλά όχι να τις καταργήσουμε εντελώς. Και στο άρθρο 18 θα μπορούσε να τροποποιηθεί κάτι όπως αναγνωρίσετε και στο έγγραφο στο Συμβούλιο. Στο άρθρο 13 και 15 στην Οδηγία για την Μεταμόσχευση Οργάνων τίθεται το θέμα της αρχής ε, της ε, δωρεάν οικειοθελούς δωρεάς και θέλουμε να υποστηρίξουμε τη γραμμή της Επιτροπής. Ήταν και πάντοτε η θέση του Κοινοβουλίου αυτή. Και εμείς έχουμε μια νομική υπηρεσία και η Επιτροπή έχει νομική υπηρεσία και κατέληξαν οι νομικέ μα υπηρεσίε σε διαφορετικό αποτέλεσμα από ότι η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου. Και βέβαια θα πρέπει ε, να ρυθμίσουμε αυτά τα οποία θέλουμε, δεν θα το αφήσουμε πλήρω στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, θα το εξετάσουμε με κριτικό πνεύμα. Η νομική υπηρεσία έχει μια πιο τεχνοκρατική εικόνα σχετικά με την προστασία ε, των δεδομένων του δωρητού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η οδηγία θα είναι επιτυχημένη αν επιτύχει η μεταμόσχευση αλλά αποβιώσει ο δωρητής. Επομένως η προστασία του δωρητού είναι ένα συγκεκριμένο σοβαρό θέμα. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εξετάσετε τη γραμμή της Επιτροπής και τις θέσεις των εμπειρογνωμόνων σας επ' αυτού. Θέλουμε μια Ευρώπη ε, ισχυρή. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξετε τη θέση σας σε αυτό το θέμα για να μπορέσετε να έχετε μεγαλύτερη επιτυχία στην Προεδρία σας. Τέλος, για το πακέτο των ε, φαρμάκων, ε, έχουμε διαφορετική άποψη στο θέμα των πληροφοριών προς τους ασθενείς. Θέλουμε όμως να είμαστε επικοδομητικοί εμείς από πλευράς Κοινοβουλίου και θέλουμε ε, να φροντίσουμε να ενημερώνονται καλύτερα οι ασθενείς. Αυτό είναι το σκεπτικό μας. Δεν θέλουμε απλώς να είμαστε αρνητικοί σε σχέση με την πρότασή σας. Θα τα παρουσιάσουμε όλα αυτά όμως, θα τα θέσουμε επιτάπητος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και ε, να σας συγχαρώ και για τις γνώσεις των Ισπανικών σας. Ε, η Ντάγμα Ροτ την επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ κυρία Χιμένε. Πολύ προσεκτικά σας άκουσα και μου άρεσε αυτό που είπατε. Ότι θέλετε να εξασφαλίσετε τη φροντίδα με υψηλή ποιότητα σε έναν κοινό χώρο υγείας στην Ευρώπη που θα σέβεται τις αρχές και τις αξίες των συστημάτων μας, παράλληλα με τις ανάγκες των ασθενών. Και επίσης θέλετε να καταργήσετε τις διακρίσεις εναντί των ασθενών. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά που είπατε. Έχει αλλάξει όμως τώρα ο ρόλος σας, γιατί μέχρι τώρα ήσασταν ένα από τα μέλη των 27 κρατών μελών. Τώρα όμως είστε η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου και τώρα πρέπει, όπως γνωρίζετε, να είστε μια πραγματική μεσάζων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πολλά θέματα η Ισπανία ακολουθούσε μία θέση στο Συμβούλιο των Υπουργών και το ανέφερε και ο κύριος Λίζες αυτά που είπε, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει η Ισπανία κατά τον ίδιο τρόπο τώρα ως Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Ε, να αναφερθώ σε κάποια θέματα στα οποία η Ισπανία δεν βρίσκεται στην κορυφή. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει το θέμα της μεταμόσχευσης οργάνων όπου είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα της Ισπανίας, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς το θέμα των υπηρεσιών υγείας διαμεθοριακά, παραδείγματο χάρη, τον έφερε και ο πρόεδρος ότι είναι μία από τις προτεραιότητε, και θα θέλαμε και εμείς να ακούσουμε από εσά, τι έχετε να μας πείτε. Θέλουμε να ακούσουμε αν το έχετε στην ημερήσια διάταξη Τη προεδρία σα. Τον Απρίλιο του 2009 έγινε η πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο, δηλαδή πάει ένας χρόνος σχεδόν. Και ξέρετε ποια είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Λέει σαφώ ότι οι ασθενείς έχουν ε, το δικαίωμα να έχουν ελεύθερη ε, μετακίνηση, ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω τα πορτοκάλια, όπω τα προϊόντα, τα υπόλοιπα. Είπατε, μιλήσατε και το έχω σημειώσει, κοινό χώρο υγείας. Πολύ καλά το είπατε. Θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τα θέματα λεπτομεριών βέβαια. Καταλαβαίνω ότι προέρχεστε ε, από μια χώρα όπου είναι διαφορετικό το σύστημα επιλογής γιατρών, παραδείγματος χάρη από ό,τι στη δική μου χώρα. Ε, τώρα όμως δεν είστε εκπρόσωπος της Ισπανίας, είστε η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Και θα ήθελα να ακούσω από εσά ε, τι θα κάνετε για τη διαμεθοριακή παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το ε, συζητήσετε ή θέλετε να το αποθήσετε και να μην το θέσετε καθόλου επιτάπητος. Ευχαριστώ πολύ σαφές ερώτημα για ένα πολύ σημαντικό θέμα και πολλές συζητήσεις έχουν γίνει στο Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Θα πρέπει να περιμένουμε από το Συμβούλιο να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Αντώνια Παρανόβα. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια, κύριε Υπουργέ. Ήταν εξαιρετική παρουσίαση των προτεραιοτήτων σας. Και είμαι βέβαιο ότι με τις επαγγελματικές σας ικανότητες και τις φιλοδοξίες σας θα καταφέρετε να επηρεάσετε τον επίτροπο, τον ή την επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία. Όμως, εδώ παλεύουμε εδώ και χρόνια με την επικουρικότητα και την αρχή αυτή στον τομέα της υγείας. Γνωρίζουμε ότι είναι πολλέ ανάγκε των ασθενών και εσεί ξεκινήσατε με μια σειρά από ευαίσθητα θέματα όπω την πρόσβαση σε καλέ και αξιόπιστε υπηρεσίε, την κλινική παρακολούθηση. Από τη δική μα την εμπειρία σε αυτό το σώμα γνωρίζουμε ότι όταν κανεί πρέπει να αγωνιστεί με το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη τα πράγματα είναι δύσκολα. Ξέρουμε ότι προσπαθούν να προστατεύσουν τα εθνικά του συστήματα πάνω απ' όλα. Και σε αντίθεση με τις, τις των ίδιων των ασθενών κάποιε φορές. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς σκοπεύετε στην πράξη να πείσετε τους συναδέλφους σας, του Υπουργού Υγεία των άλλων κρατών μελών, τουλάχιστον να περάσει η οδηγία για την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Και εσείς τι νομοθέτημα θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα προωθούσε την ασφάλεια και την ποιότητα διασυνοριακά. Έχετε ήδη προχωρήσει σε τίποτε διαπραγματεύσεις, προκαταρκτικές συνομιλίες. διότι θα πρέπει να πετύχετε τη στήριξη της Βελγικής και της επόμενης Προεδρίας για να είσαστε βέβαιοι ότι θα πετύχετε. Εδώ έχετε ένα εξάμεινο μπροστά σας. Θα πρέπει να μας πείτε τι θεωρείτε ότι είναι εφικτό από το φιλόδοξο πρόγραμμα που έχετε θέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ, για την εξαιρετική σας ε, παρουσίαση. Τρία πράγματα με ανησυχούν κυρίως. Πρώτα απ' όλα, η ε, ενίσχυση της διαφάνειας σε ζητήματα της πληροφόρησης για τις παρενέργειες ε, στα συσκευασίες των φαρμάκων και στα πλαίσια του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνηση. Είναι σημαντικό αυτό σήμερα γιατί γνωρίζουμε ότι οι ασθενεί δυσκολεύονται τη σημερινή μέρα να αποκτήσουν ε, αξιόπιστες πληροφορίες, να έχουν στα χέρια του αξιόπιστες πληροφορίες για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Επίση, ποιε οι επαφέ σα με τα Υπουργεία υγεία και τα Υπουργεία περιβάλλοντο. Πώ θα διασυνδεθούν αυτά μεταξύ του. Υπάρχουν πάρα πολλέ χώρε που δεν είναι ικανοποιημένε από τον ορισμό των ε, επικίνδυνων ουσιών λόγου χάρη. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε κάποια πράγματα να τα αποσαφηνίσουμε, ιδίω ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τη σχέση του με τα φάρμακα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποιε συγκεκριμένε διαδικασίε για την αδειοδότηση. Όπω ξέρετε, υπάρχει ένα άρεκτο δεσμό μεταξύ περιβάλλοντο και υγεία ε, Πολλέ φορέ ο επίτροπο που είναι φορτισμένος με τα θέματα βιομηχανία, έχει την τάση λόγω χάρη όλα να τα αναμειγνύει. Όμω, εδώ θέλουμε να πετύχουμε να έχουμε έναν υγιή πληθυσμό στην Ευρώπη. Αυτό μα ενδιαφέρει. Οι Υπουργοί λοιπόν Υγεία θα πρέπει να συνεργαστούν με τον αρμόδιο Επίτροπο για να καταλήξουν σε κάτι συγκεκριμένο. Περιμέναμε λοιπόν πολύ για να δούμε συγκεκριμένα αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα. Θα πρέπει να γίνουν κατάλληλε διασυνδέσει μεταξύ υγεία, περιβάλλοντο και βιομηχανία. Επίση, μιλήσατε για τη στρατηγική καταπολέμηση τη υπερκατανάλωση αλάτων και ε, αλατιού. Θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό μα ενδιαφέρει πολύ και στο Κοινοβούλιο. Μελετώντας τα σχετικά προγράμματα, καταλάβαμε ότι αυτό είναι το καταλληλότερο πρόγραμμα για να καταπολεμήσουμε τις καρδιοαγγειακές παθήσεις. Το Κοινοβούλιο λοιπόν θέλει να γνωρίζει εάν θα επαναφέρεται το θέμα αυτό στο Συμβούλιο ή όχι. Κυρία Μαρίζα Ματία, στην επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, καλώ ήρθατε κυρία Υπουργέ. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση άκουσα την παρουσίασή σα και τα λόγια σα. Νομίζω ότι θέσατε τους βασικούς προσανατολισμούς της Προεδρίας σας και πολύ καλά αναφερθήκατε στους φορείς υγείας και το πόσο έμφαση θα του δώσετε κατά τη διάρκεια τη θητεία σα. Θέλω να θέσω τώρα κάποιε ερωτήσει. Αναφέρατε ω μια από τι προτεραιότητε ε, τη Προεδρία σα να προχωρήσετε στο πακέτο σε σχέση με τα φάρμακα και ιδίω σε σχέση με τα ψευδεπίγραφα φάρμακα και την φαρμακοεπαγρύπνηση. Επειδή είμαι εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα συγκεκριμένα, και ήδη ξεκινήσαμε τις συζητήσεις με προσώπους της κυβέρνησής σας, υπάρχει ένα σημείο που δεν ήταν πολύ σαφής η τοποθέτηση του Συμβουλίου εδώ. Και μάλιστα ευθύς εξ αρχή. Κυρία Υπουργέ, εσείς μπορείτε να μας δώσετε κάποια περαιτέρω πληροφορία για το θέμα αυτό. Συμπερίληψη ή όχι των πωλήσεων φαρμάκων και ψευδεπίγραφων φαρμάκων στο διαδίκτυο. Πωλήσει στο ίντερνετ λοιπόν είναι μια από τις βασικές ε, διόδους των ψευδεπίγραφων φαρμάκων στην αγορά. Είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε αυτό στην κοινή γνώμη αν δεν συμπεριληφθεί. Και αυτό ακριβώς ήθελα να μου πείτε. Και ένα ακόμη ερώτημα. Δώσατε μεγάλη έμφαση στις ε, χρόνες παθήσεις, στις σχέσεις με τη διάρκεια ζωής, στην υγεία του πληθυσμού. Υπάρχει μια χρόνια πάθηση που δεν έχει απαραίτητα σχέση με την αύξηση του προσδόκιμου ζωή και πολύ συχνά την παραμελούμε. Είναι ο διαβήτη. Θα ήθελα λοιπόν να δώσετε κάποια έμφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε αυτή την ε, πάθηση. Πλήττει ένα μεγάλο μέρο του πληθυσμού και υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που δεν έχουν συγκεκριμένε πολιτικέ ούτε για να την ε, προλάβουν ούτε για να την καταπολεμήσουν την ασθένεια αυτή. Φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει και άλλου βουλευτέ και ήθελα να ξέρω αν έχετε προγραμματίσει κάποια βήματα για του επόμενου μήνε προ αυτή την κατεύθυνση. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα ζήτημα το οποίο μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές προσωπικά, διότι είμαι συγγήτρια για την οδηγία σε σχέση με τις διασυνοριακέ υπηρεσίες υγείας. Πολλοί από τους συναδέλφους μου γνωρίζουν ότι έχουμε συζητήσει για τα θέματα αυτά. Εδώ έχει παίξει πολύ αρνητικό ρόλο η Ισπανία όμως. Το Δεκέμβριο και εφόσον εσείς εξτατεύσατε κατά της οδηγίας αυτής, προσπαθήσατε να πείσετε κράτη-μέλη να σας ακολουθήσουν. Και αυτό ουσιαστικά οδήγησε στο να αναβαγίσουν οι συζητήσεις και η συμφωνία που περιβαίναμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία όπως φαντάζεστε. Προηγουμένως στην παρέμβασή σας είπατε ότι θα αποσπάσετε συνένεση για την οδηγία. Ναι, εγώ να σας πω διερωτώμεθα πώς θα αποσπάσετε συνένεση ενώ εξτατεύσετε κατά της οδηγίας αυτής και μάλιστα χωρίς καθόλου να κρυφτείτε, απροκάλυπτα. Τώρα πώς θα σε εμπιστευτούμε, μας λέτε ότι θα επιδιώξουμε συνένεση. Ε, για ε, διευκρινίστε το κάπω αν μπορείτε, διότι ο συνάδελφο πολύ σωστά το θύμισε, σε αυτή την οδηγία εμεί είχαμε μια τοποθέτηση για τους εξελαχίστων κανόνε. Θέλαμε απλώ να παραμείνουμε σε όσα ορίζουν οι αποφάσει του ΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν ζητούσαμε περισσότερα. Αυτό που θέλαμε εμεί από το Κοινοβούλιο είναι εμεί οι νομοθέτε και όχι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να διευθετεί αυτά τα θέματα. Ήμασταν αρκετά λογικοί και μετρημένοι και προτείναμε κάτι στην οδηγία αυτή που να είναι όσο το δυνατόν αντικείμενο συνένεση, εφόσον λαμβάνει υπόψη τις αποφάσει του δικαστηρίου και εσεί τον μπλοκάρατε. Πείτε μας λοιπόν πείτε μας τι σκοπεύετε να κάνετε, αλλά συγκεκριμένα. Δεν θέλουμε εδώ λόγια και πομπόδι, αλλά να μας πείτε συγκεκριμένα τι θα κάνετε για να αναβιώσει αυτό το κείμενο. Διότι σήμερα φαίνεται ότι είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε τη Βελγική Προεδρία. Για να αρχίσουμε να ελπίζουμε να προχωρήσει το κείμενο αυτό, το οποίο είναι σημαντικό όχι μόνο για το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά για όλους τους ασθενείς στην Ευρώπη. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Ο Αντρέ Περίγιον θα είναι επόμενο ομιλητή και μετά θα δώσουμε το λόγο στην Υπουργό να απαντήσει στον πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σαφήνεια, για την ακρίβεια της ε, παρουσίασής σας και πραγματικά σας παρακινώ ε, να συνεχίσετε με την ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο να αναφέρεται δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά είναι και μέσο για να υπάρχει ισότητα μεταξύ όλων. Αναφερθήκατε σε πολύ σημαντικά θέματα, μεταξύ αυτών και τη μεταμόσχευση οργάνων και αναφερθήκατε και στη σημασία ε, του πλαισίου υγείας. Ε, θα ήθελα να σταθώ σε δύο πράγματα. Ε, το πρώτο είναι μια προσωπική άποψη. Η ιδέα του να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα για τη μεταμόσχευση οργάνων, για τους δωρητές οργάνων, τι πιστεύετε ότι μπορείτε να γίνεται. Και επίσης, αναφερθήκατε και στο δίκτυο το ευρωπαϊκό και επειδή είναι πολύ σημαντικό, και μας είπατε και ποιες θα είναι οι προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας για τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι γίνεται από αυτού. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας γιατί ήσασταν πολύ ακριβείς και πολύ σαφείς. Πολλές ερωτήσεις. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι για τις ερωτήσεις σας. Καταρχάς θα ήθελα να κάνω μια γενική διευκρίνηση. Η Ισπανία είναι η Προεδρία. Είναι η Προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει συνειδητοποιήσει πλήρως το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει ε, και ε, θέλει να ε, είναι ο διαμεσολαβητής για όλες τις χώρες μέλη και είναι πάρα πολύ σαφές και ποια είναι η θέση μας σε κάθε στιγμή. Και ελπίζω να σας δώσει ευκαιρία να το αποδείξουμε αυτό ε, στη διάρκεια των εργασιών μα. Ναι, μεν θέλουμε να τηρήσουμε τη βούληση όλων των κρατών μελών, αλλά εργαζόμαστε ώστε να προχωρήσουμε όλε τι πρωτοβουλίε με τον τρίο των προεδιών, δηλαδή με το Βέλγιο και την Ουγγαρία, αλλά και με τι υπόλοιπε χώρε μέλη στα διάφορα συμβούλια και σε επίπεδα συντονισμού στα οποία πρέπει να καθορίσουμε τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Δεύτερον, και θα απαντήσω και σε κάποιες ερωτήσεις που μου ε, έγιναν όσον αφορά στην ε, οδηγία για τη διαμεθοριακή περίθαλψη. Όταν σα είπα στην αρχική μου παρέμβαση ότι θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, είναι γιατί πραγματικά θα δουλέψουμε για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Η Ισπανία προάσπισε τη θέση της στεναρά. Δεν ήταν κατά της οδηγία εν γέννη, ήταν υπέρ κάποιων αρχών τι οποίε θεωρούμε βασικές και αυτή είναι ότι η υγεία είναι δημόσιο αγαθό, είναι δημόσια υπηρεσία, δεν είναι ένα επιπλέον ε, ε, σημείο εμπορίου. Και γι' αυτό για μας ήταν θεμελιώδες να διασφαλίσουμε καταρχάς την ασφάλεια των ασθενών και δεύτερον την ποιότητα της διαμεθοριακής περίθαλψης. Που τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ζητήσαμε να υπάρχει πρώτερη έγκριση για να υπάρχει μια υπηρεσία περίθελψης ώστε κάποιος να μπορεί να επιλέξει για ιατρικούς λόγους και δεύτερον για να διασφαλίσουμε την ποιότητα της περιθέψης. Θέλουμε λοιπόν ο χώρος τον ο οποίος επιλέγεται να βρίσκεται εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δηλαδή να είναι ένα δημόσιο ε, κέντρο ή ένα πιστοποιημένο κέντρο υγείας. Και έτσι προσπαθούμε να ρυθμίσουμε κάτι το οποίο μας φαίνεται θεμελιώδες. Ζητήσαμε περισσότερη φιλοδοξία, διότι μας φάνηκε ότι αυτό το οποίο παρουσίασε το Συμβούλιο και δεν ήταν αρκετό και μάλιστα επειδή δεν υπήρχε ομοφωνία ε, θεωρούμε ότι πρόκειται για κάτι το οποίο εξακολουθεί να μην ρυθμίζεται στους κανόνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή για τα συστήματα ε, κοινωνικής ασφάλισης. Είμαστε πεπισμένοι και φιλόδοξοι και θα σας το αποδείξουμε. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όπως πάντα εργαστήκαμε με επικοδομητικό πλεύμα, με πνεύμα συνεργασίας και κυρίως με μια φιλοδοξία η οποία είναι να είμαστε στην υπηρεσία του πολίτη. Ποιότητα και ασφάλεια. Επιμένω σε αυτό γιατί θεωρούμε ότι η υγεία δεν είναι επιπλέον αγαθό, είναι μια δημόσια υπηρεσία. Και με αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και θα γνωρίζουμε και την άποψη του νέου Επιτρόπου με τον οποίο έχω προβλέψει να συναντηθώ. Όσον αφορά τώρα στην οδηγία για τη μεταμόσχευση ε, οργάνων. Είμαστε υπέρ της δωρεάν μεταμόσχευσης και είμαστε και υπέρ της προστασίας του δωρητή. Στην πρόταση του Συμβουλίου λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ένα μοντέλο δωρεά το οποίο θα είναι αλτρουιστικό και θα προστατεύεται ο δωρητής. Έχουν γίνει πάρα πολλέ πρόοδοι στο θέμα αυτό. Ε, υπήρξε πάρα πολύ σημαντική, εξαιρετική δουλειά και είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε επί τη βάση της ποιότητας, της προστασίας και κυρίως με το στόχο ε, της ισότητας. Όσον αφορά τώρα το θέμα των φαρμάκων. Είναι σαφές ότι στο θέμα των φαρμάκων έχουμε μια πολύ σημαντική πρόοδο όσον αφορά σε ψευδεπίγραφα ε, φάρμακα και στη φαρμακοεπαγρύπνηση. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε συμφωνία σε θέματα πληροφόρησης, ενημέρωσης του καταναλωτή, του ασθενούς. Γι' αυτό ακριβώς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όπως κάναμε για τις δύο αυτές οδηγίες, για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα και για τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Θεωρούμε ότι εδώ έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε, έχουν γίνει σημαντικά βήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα και αξίζει τον κόπο να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Διαφάνεια στη φαρμακοεπιγρύπνηση. Συμφωνούμε. Θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια για τους πολίτες σε σχέση με τους δυνητικούς κινδύνους των φαρμάκων. Οτιδήποτε προσδίδει περισσότερη ασφάλεια στον ασθενή, περισσότερη ασφάλεια στον καταναλωτή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τώρα ε, στην οδηγία για το αλάτι, να σας πω ότι εργαζόμαστε, να σας πω ότι σήμερα έγινε και μια συνεδρίαση με την οποία ε, καταλήξαμε σε συμφωνία, ε, εκπρεμούν κάποια μικροθέματα και επομένως θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε στο Συμβούλιο του Ιουνίου αυτή την πρωτοβουλία όσον αφορά στη μείωση της περιεκτικότητας σε αλάτι κάποιων φαρμάκων και την ε, πρόληψη των καρδιαγκιακών παθήσεων. Όσον αφορά τη διατροφική ασφάλεια, θα ακούσουμε τι έχει να μας πει το πάνελ της ΕΦΣΑ και θα λάβουμε υπόψη το θέμα της, ε, ε, της Βουλής της ΕΦΣΑ για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Και να σας πω και κάτι για το eHealth. Ε, θα προχωρήσουμε τις ε, προτάσεις της Σουηδικής ε, Προεδρίας για το θέμα αυτό. Θα προτείνουμε νέες συμφωνίες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την ψηφιακή ιατρική ε, στην κοινοτική πολιτική και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ιατρική περίθαλψη προς αυτό το χώρο. Γι' αυτό λοιπόν θα προχωρήσουμε την πολιτική και στρατηγική ε, δέσμευση, θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών και ασθενών και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μεγαλύτερη νομική ασφάλεια και σαφήνεια για την προστασία των δεδομένων. Πρόκειται για μια πολιτική υγείας, ψηφιακής υγείας, η οποία θα περιλαμβάνεται στην ατζέντα ε, για μετά το 2010 και φυσικά θα ε, προσπαθήσουμε να τις δώσουμε και τη δέουσα θέση στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Στη Βαρκελόνη θα γίνει και η υπουργική διάσκεψη με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συζητήσουμε το e-health for health και e-health ε, για να έχουμε βιώσιμη περίθαλψη. στο σύστημα υγείας έχουμε μια γυροάσκουσα κοινωνία, μια κοινωνία που γυράσκει πάρα πολύ γρήγορα και ταυτόχρονα ε, επειδή αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής και έχουμε και μείωση του ποσοστό θνησιμότητας, αυξάνονται οι χρόνιες παθήσεις. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν το e-health θεωρούμε ότι θα μπορέσει να συνεισφέρει πολύ θετικά και θα μπορέσουμε να έχουμε πιο αποδοτικά συστήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Και η Ισπανία λοιπόν θα είναι μία από τις ε, χώρες που θα ακολουθήσουμε ηγετική στάση σε αυτά τα θέματα της διαμεθοριακής περιθέλψης. Και σίγουρα πολλοί από τους ευρωβουλευτές χαίρονται ιδιαίτερα για τη θέση σας αυτή. Η κυρία Βέσλουν την επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη ικανοποίηση να βλέπουμε ότι θα δώσετε έμφαση στα θέματα της κινητικότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Αλλά είναι κάπως κρίμα να βλέπει κανείς ότι υπάρχει ανισότητα στην υγειονομική περίθαλψη και ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που παραμένει σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε το καταλληλότερο σύστημα για να αποφύγουμε ακριβώς τις ε, καταστάσεις ε, ανισότητας. Έχω εδώ να σας θέσω ένα ερώτημα. Όχι τόσο πολύ για την ισότητα. Ένα πρώτο ερώτημα για την πληροφόρησή μας για τα τρόφιμα. Στο Συμβούλιο των Υπουργών πώς έχουν προχωρήσει οι σχετικές συζητήσεις. Υπάρχει συμφωνία σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις για τα θρεπτικά συστατικά λόγου χάρη. Υπάρχουν ακόμη σημαντικά ζητήματα που εκκρεμούν αλλά ενδεχομένω σύντομα να επιληθούν. Υπάρχουν σοβαρές αποκλήσεις απόψεων. Κατά την άποψή σα πότε θα μπορέσουμε κατά πάσα πιθανότητα να περιμένουμε μια απόφαση. Πού βρίσκεστε στο Συμβούλιο των Υπουργών σχετικά. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Αυτό που μας είπατε για τη μικροβιολογική αντεκτικότητα. Εδώ ξέρετε ότι υπάρχει θέμα με τα εμβόλια στην Ευρώπη και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Θα σκύψετε στο θέμα αυτό επί Ισπανικής Προεδρίας. θα εξετάσετε τη χρήση των αντιβιωτικών και την ανθεκτικότητα που δημιουργείται απέναντι στα μικρόβια και στα αντιβιωτικά μάλλον στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο ή να κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Να... Θα συμπεριλαμβάνω όλους. Ελιζαμπέτα Βουκασιέφκα. Ευχαριστώ, Υπουργέ, για την παρουσίασή σας. Αλλά πρέπει να πω ότι εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει καμιά χώρα που θα μπορούσε κάνει ως προς τη δημόσια υγεία της να περιγραφεί ως ιδεατός τόπος. Χαίρομαι που ακούω ότι σε ό,τι αφορά τις μεταμοσχεύσεις η Ισπανία εδώ βρίσκεται στην πρωτοπορία. Κάποιες χώρες ακόμη παλεύουν με το πρόβλημα της έλλειψης δωρητών. Το να υπάρχουν άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να δωρήσουν τα οργανά τους είναι ήδη σημαντικό. Μπορείτε λοιπόν να μοιραστείτε μαζί μας τις απόψεις σας για το ενδεχόμενο να γίνει εξτατεία ευαισθητοποίησης, να ενθαρρύνουμε το κοινό να δωρίζει τα όργανα. Και βλέπω ότι το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε ξανά βάσει τη ημερήσια διαταξή μα σήμερα. Όμω, εγώ θέλω να ακούσω και τι δικέ σα απόψει. Και για το εμβόλιο τη γρήπη του ιού H1N1. Σε σύγκριση με τι τεράστιε δαπανέ που έγιναν από τα κρατη το μόνο που μπορεί κανεί να κάνει είναι να ρωτηθεί αν τελικά σωστά δαπανίσαμε αυτά τα χρήματα προ αυτή την κατεύθυνση ή θα πρέπει να τα έχουμε διοχετεύσει σε άλλου τομεί τη ε, δημόσια υγεία. Για την διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών υγεία, θα έλεγα ότι η κυρία Γκροστέτ μου έκλεψε λιγάκι την έμπνευση. Η Ισπανία είναι μια από εκείνε τι χώρε που μπλόκαραν την ε, πρόθεση τη οδηγία. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η οδηγία ώστε να είναι αρκετά φιλόδοξη από τη δική σας τουλάχιστον προοπτική. Γνωρίζουμε ότι το σύστημα υγείας των 27 κρατών μελών είναι πολύ διαφορετικό από τη μια χώρα στην άλλη. Θα ήθελα η Πολωνία ασθενής να έχουν δικαίωμα να λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλες χώρες. Όμως τα συστήματά μας έχουν περιορισμένους πόρους και δυναμικό. Πρέπει λοιπόν να μας πείτε κάτι λίγο πιο σαφές ως προς αυτό. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας τέθησαν ε, πολλά ξεκάθαρα ερωτήματα και από όλες τις πολιτικές ομάδες. Μου κάνει εντύπωση ότι το Συμβούλιο δεν είναι έτοιμο να εφαρμόσει αυτά τα οποία έχει ζητήσει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και αυτό μας αφορά ιδιαίτερα στο θέμα της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών υγείας. Λέτε ότι είστε όντως ε, ειλικρινείς μεσάζων, αλλά για το θέμα των φιλοδοξιών δεν ξέρουμε πόσο μακριά θέλετε να προχωρήσετε. Θα μπορούσατε να μας πείτε πού βρίσκονται οι φιλοδοξίες σας. Μπορεί να έχετε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, αλλά πολύ συγκεκριμένα. Τι θα κάνετε πού θέλετε να δώσετε μεγαλύτερη σημασία στην ευρωπαϊκή διάσταση αυτού του θέματος. Όλοι είμαστε υπέρ του ε, ε, καλού ε, των ασθενών, αλλά οι ασθενείς έχουν μεγάλες δυσκολίες όταν θέλουν διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας. Μπορεί να είναι για το καλό τους, αλλά δεν το βλέπουν στην πράξη. Είπατε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ νοσοκομείων στα κράτη-μέλη. Και στο θέμα της αντιμετώπισης λιμωδών νόσων, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Γιατί να μην έχουμε όμως ένα ελάχιστο επίπεδο, υπό την έννοια του name and shame, δηλαδή να κατονομάσουμε και να κατηγορήσουμε αυτούς οι οποίοι δεν προσφέρουν επαρκώς ποιοτικέ υπηρεσίες. Να έχουμε δηλαδή ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας και να πούμε ότι για μας τους Ευρωπαίους αυτό είναι ένα ελάχιστο πρότυπο και όποιος δεν το επιτυγχάνει θα πρέπει να το γνωρίζουν και οι ασθενείς, να τους κατονομάσουμε δηλαδή αυτό αυτούς που δεν ε, έχουν επαρκή ποιοτικά πρότυπα. Ένα τρίτο ερώτημα που αναφέρθηκε και η συνάδελφος Λουκασένθηκα σε αυτό. Ε, μιλάμε για την καταπολέμηση της ε, πανδημίας της γρήπης. Ε, στη Γερμανία αγοράσαμε 40 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων παραπάνω από αυτό που χρειαζόμασταν. Ε, ε, θα έπρεπε να υπάρχει κάποια αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή ε, να παραγγέλναμε από κοινού μια ποσότητα εμβολίων και να μπορούσαν να εφοδιαστούν τα κράτη-μέλη με τα φάρμακα τα οποία χρειάζονται εκεί όπου τα χρειάζονται. Ενώ καταφεύγουμε με μεμονωμένες λύσεις σε κράτη-μέλη και αυτό οδηγεί σε τεράστιο κόστος ενώ θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τους πόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Wenn Ίσως αν τα παράγγελνε η Ευρώπη και παράγγελνε 300 εκατομμύρια, μπορεί πάλι να είχαμε ξεπεράσει τις απαραίτητες ποσότητες εμβολίων. Ο Στρεμόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σε πρόσφατη... σε πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος αναφέρεται ότι οι, οι διαδικασίες έγκρισης των πωλήσεων, οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση των φαρμακευτικών ε, προϊόντων πρέπει να παίρνουν υπόψη και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Τα φαρμακευτικά προϊόντα θα πρέπει να κατατάσσονται, λέει ακόμη, ανάλογα με τους κινδύνους που έχουν για το περιβάλλον. Ποια είναι η γνώμη σας. Μέσω της φαρμακοεπαγρύπνησης ε, θα πρέπει να παρακολουθούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τι προγραμματίζεται γι' αυτό. Επίσης, είπατε ότι θα ακούσετε για τα γενετικά τροποποιημένα την ε, άποψη της ΕΦΣΑ. Εδώ σε αυτή την αίθουσα ο υποψήφιος Επίτροπος Υγείας είπε τουλάχιστον ότι θα το μελετήσει. Και ιδιαίτερα μάλιστα εφόσον η ΕΦΣΑ είναι αμφιλεγόμενος οργανισμός και όσον αφορά τουλάχιστον τις σχέσεις των στελεχών, κάποιων στελεχών της με τις εταιρείες βιοτεχνολογίας. Θα πρέπει να μας πείτε από τη στιγμή που στην Ισπανία καλλιεργείται το καλαμπόκι μόν 810 εδώ και 10 χρόνια. Και έχει αποδειχθεί ότι, από έρευνα ότι μια τοξίνη έχει αυξήσει την τοξικότητα των εδαφών και των γεωσκολίκων με επιπτώσεις στις καλλιέργειες, στα έντομα και τις πεταλούδες. Έχετε υπόψη σας έρευνα ή εν πάση γενικότερα για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία. Με δεδομένο ότι το καλαμπόκι μόνο 810 χρησιμοποιείται και για τις ζωοτροφές, ρωτώ αν έχετε υπόψη σας κάποια έρευνα για επιπτώσεις στη διατροφική ασφάλεια. Και τέλος, Εφόσον συζητάμε και για τη γρήπη είτε ένα ή ένα, ε, πώς, ε, πώς αξοδέψατε ακριβώς την Ισπανία εσείς για τα εμβόλια και αν συμφωνείτε με την άποψη ότι ήταν ένας σχεδιασμένος πανικός χωρίς, που κόστησε χωρίς σοβαρό λόγο. Äh, η Υπουργό είναι τώρα Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Δεν κάθεται εδώ ανάμεσά μα ω Ισπανή Υπουργό. Είναι η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Πιλάρα Γιούζο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την ε, παρουσίασή σα και το πρόγραμμά σα, ε, για το οποίο δεν έχω καμία ένσταση. Φαίνεται καταπληκτικό και πολύ φιλόδοξο. Έχω κάποια σχόλια όμως και ερωτήσεις για το θέμα το οποίο προέκυψε αρκετές φορές την διαμεθοριακή ιατρική περίθελψη και την κινητικότητα των ασθενών. Στη θεωρία όλοι συμφωνούμε. Πρέπει να υπάρχουν ε, παροχές ποιότητας, είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να γίνει είναι μεν δημόσιο αγαθό, αλλά δεν είναι δωρεάν. Και με όλες τις, ε, τους ιατρικούς συλλόγους με τους οποίους συνάντησα, διότι με αφορά το θέμα, η απόφαση είναι ομόφωνη. Ναι μεν, αλλά σε όλες τις χώρες δεν έχουμε τις ίδιες ε, παροχές θέλψη τα ίδια νοσοκομεία, επομένως ασθενής κοιτάει να δει πού θα του προσφέρουν καλύτερη περίθελψη. Αλλά μετά πώς αποζημιώνονται αυτές οι δαπάνες. Και φυσικά δεν θέλω καν να αναφέρω τι σημαίνουν αυτές οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία. Στην Ισπανία έχουμε πάρα πολλά τέτοια, τέτοιες επιπλέον δαπάνες λόγω του αυξημένου αριθμού ε, τουριστών που έχουμε. Αλλά πραγματικά αυτό ενδιαφέρει τους ιατρικούς συλλόγους. Ποιος θα ε, καταβάλει τις δαπάνες για όλες αυτές τις ε, διαμεθοριακές ε, παροχές υγείας. Επίσης, το θέμα της διατροφικής ασφάλειας. Εδώ στην Ευρώπη είμαστε πάρα πολύ φιλόδοξοι. Έχουμε κανόνες πολύ ε, υψηλής ε, ποιότητας ε, ασφάλειας τροφίμων και το ίδιο περιμένουν και από εμάς οι καταναλωτές μας. Σε γενικές γραμμές η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων είναι σχετικά καλή. Αλλά εισάγουμε προϊόντα, κυρίως γεωργικά προϊόντα από τρίτες χώρες που δεν τηρούν τους ίδιους κανόνες και φυσικά δεν μπορούμε να αποφύγουμε την εισαγωγή τους. Δεν μπορούμε να την αποφύγουμε διότι ο ΠΟΕ το απαγορεύει. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αναζητήσουμε κάποιο μηχανισμό για να επιλύσουμε το πρόβλημα. Παραδείγματο χάρη, οι ΗΠΑ έχουν επιθεωρητέ. Εμεί έχουμε ε, στην Ισπανία Αμερικανού επιθεωρητέ, οι οποίοι έρχονται εδώ και έρχονται στην Ισπανία και ελέγχουν πώ ε, παρασκευάζεται το διάσημο χαμόνι μπέρικο. Αλλιώ δεν μπορούμε να του εξάγουμε στην, ε, τι θα κάνουμε εμείς λοιπόν για να ελέγξουμε την κατάσταση, γιατί εμείς επιβαρύνουμε τους παραγωγούς μας με δαπάνες τις οποίες δεν έχουν οι άλλοι και φυσικά δεν μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικοί. Επιπλέον, με τους νέους κανονισμούς για τα φυτοφάρμακα, στη Κανάρια νησιά δεν θα μπορέσουμε να ψεκάζουμε για την άσπρη μύγα και φυσικά δεν θα πρέπει να εισάγουμε προϊόντα τα οποία ε, στα... παράγονται στα Κανάρια νησιά και ε, δεν θα μπορούμε πλέον να τα παράγουμε γιατί θα απαγορεύεται ο ψεκασμός. Τίποτα άλλο, θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για τις προτεραιότητες που αναφέρατε. Τα θέματα υγείας είναι θέματα που είναι ιδιαίτερα προσφυλή και για μας, αλλά και στους πολίτες της Ευρώπης γενικότερα. Ο κύριος ε, Νταλή, ε, υποψήφιος επίτροπος, ε, κατά την ακρόαση, ανέφερε το θέμα της πληροφόρησης και ανέφερε ότι χρειάζεται υψηλότερη προστασία των ασθενών. Τι συμπληρωματικά μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν στον τομέα της φάρμακοεπαγρύπνησης για να προστατεύονται καλύτερα τα δικαιώματα των ασθενών. Ευχαριστώ. Μισελ Ριβαζή, τελευταία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, κυρία Υπουργέ. Ήθελα να σταθώ στα θέματα υγείας. Εάν κοιτάξει κανείς την κατάσταση της δημόσιας υγείας στην Ευρώπη, ιδιαίτερο στι βιομηχανοποιημένε χώρες, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μια επιδημία θα έλεγε κανείς, επίπεδο καρδιοαγγειακών παθήσεων και μάλιστα καρκίνο. Στη Γαλλία έχουμε 150.000 νεκρούς από καρκίνο το χρόνο. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι ανέφεραν τη γρήπη H1N1, αλλά αν δει κανεί τα δις που δαπανίσαμε στη Γαλλία, 2,2 μόνο στη Γαλλία, για 94.000 δόσεις εμβολίου, αναρωτιέμαι κι εγώ με τη σειρά μου και ήθελα να ξέρω ποια είναι η δικιά σας η απάντηση. Τι πιστεύετε για την κατασπατάληση αυτή των δημόσιων πόρων σε κάθε κράτος, ακόμα και αν κάθε κράτος ακολούθησε διαφορετική πολιτική, σε σχέση και με άλλες προτεραιότητες, οι οποίες τελικά επλήγησαν. Θα μπορούσαν όμως να τους είχαν δοθεί περισσότερα κονδύλια. Αυτό θα πρέπει να μας χρησιμεύσει ως δίδαγμα πώς θα επαναπροσανατολίσουμε την, την πολιτική αυτή ακριβώς και τι λύσεις προτείνετε εσείς για να υπάρχει μια ανεξάρτητη πολιτική. Πιο ανεξάρτητη από αυτήν που υλοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και το δεύτερο μου ερώτημα αφορά τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Ως τώρα οι οργανισμοί αυτοί δεν ήταν τομέας της αρμοδιότητάς σας. Τώρα όμως έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα του χώρου της υγείας. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με πρωτόκολλα παρακολούθησης της υγείας από τα εργαστήρια και σε σχέση με ό,τι αφορά τις συνέπειες από την κατανάλωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στην υγεία. Ένα παράδειγμα στα ποντίκια, ε, βλέπουμε ποιες είναι, οι επιπτώσεις σε εκτροφής που, στην εκτροφή ποντικών για τρεις μήνες πώ θα αλλάξουν τα πρωτόκολλα για να αυξηθεί αυτή η διάρκεια. Να μπορεί κανεί να έχει μια καλύτερη εικόνα τη επίδραση των γενετικώ τροποποιημένων στον, ε, στην υγεία και στον οργανισμό. Ευχαριστώ. Ακούσατε τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Θα δώσουμε και πάλι το λόγο στην Υπουργό που έχετε και πάλι τη δυνατότητα να απαντήσετε. Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και του αξιότιμους ευρωβουλευτέ. Ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω σε όλες σα τι Θα ξεκινήσω με την ε, ενημέρωση στον καταναλωτή για τα διατροφικά προϊόντα. Η πρόταση κανονισμού θεωρούμε ότι είναι κάτι θετικό. Πρόκειται για μία οδηγία η οποία αφενός ε, συγκεντρώνει όλα τα θέματα της ετικετοθεσίας και επίσης προσπαθεί να ρυθμίσει όλες τις ε, ασυνέπειες που έχει η φυστάμενη ε, νομοθεσία και προσπαθούμε να βρούμε και τον πιο εναρμονισμένο τρόπο για να δίνονται πληροφορίες στους καταναλωτές και επίσης υπάρχουν και κάποιες απαιτήσει σε θέματα ευθύνης για τους ε, για όλους όσους συμμετέχουν στην ε, παροχή ενός διατροφικού προϊόντος. Θεωρώ ότι είναι μια νομοθεσία ιδιαίτερο σημαντική, όχι μόνο γιατί βελτιώνει την εσωτερική αγορά, αλλά και γιατί θεωρούμε ότι θα ε, βελτιώσει την προστασία και των καταναλωτών, αλλά και από πλευράς υγείας, διότι εδώ αυξάνονται οι δυνατότητες να έχουμε μια συνειδητή επιλογή που θα γίνεται μέσω πληροφοριών οι οποίες θα είναι αποτελεσματικές και σωστές μέσω της ετικέτας, μέσω της ε, φύσης του προϊόντος και του περιεχόμενου των συστατικών προϊόντων, των συστατικών ε, ενός ε, τροφίμου αυτό το ε, νομοθετικό κείμενο το εκπώνεσε η Σουηδική Προεδρία. Εμείς προχωρούμε την πρόταση. Την έχει εξετάσει το Συμβούλιο εδώ και 1,5 χρόνο και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία σε θέματα τα οποία ε, μας ενδιαφέρουν για το θέμα αυτό. Η Ισπανική Προεδρία θα συνεχίσει τις συζητήσεις και θέλουμε να έχουμε μια πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο του Ιουνίου για την ε, πρόταση αυτή και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του θέματος. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να έχουμε μια γενική συμφωνία για την ε, πρόταση κειμένου και εδώ έχει προχωρήσει πάρα πολύ το θέμα και η ομάδα εμπειρογνωμόνων και φρονώ ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό οτιδήποτε καταφέρουμε να πετύχουμε σε αυτή την πρόταση κανονισμού. Όσον αφορά τώρα στην ε, αντιμικροβιακή εντοχή. Αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι όλα τα κράτη-μέλη προσπαθούν να δουν τι γίνεται σε θέματα ασφάλειας ασθενών και εξακολουθούμε να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό από πλευράς Ισπανικής Προεδρίας. Για τη γρήπη τώρα. Σαφώς υπάρχει συζήτηση εν εξελίξει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπάρχει συζήτηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εξακολουθεί να απασχολεί τους πολίτες. Αρκετοί ευρωβουλευτές με ρώτησαν για την γρήπη. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έζησα την επιδημία, την εμφάνιση του ιού ε, και μόλις όταν εμφανίστηκε μόλις είχαν αναλάβει καθήκοντα από δύο εβδομάδες. Όταν ε, είχαμε την κατάσταση επιφυλακής από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας λάβαμε και τον αριθμό των ε, ασθενών. Είχαμε ελάχιστα περιστατικά και από τις δύο, στις δύο ημέρες είχαμε ήδη 100 θανάτους σε ελάχιστες ημέρες. Μέσα σε δύο εβδομάδες είχαμε περιστατικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και ξαφνικά ε, σε ένα μήνα είχαμε φτάσει στις 50 χώρες. Σε ελάχιστες μέρες ε, είχαμε ήδη 62 χώρες και το επίπεδο μετάδοσης ήταν πολύ ψηλό. Θα θυμάστε όλοι τις εικόνες ε, ολόκληρων χωρών που έκλειναν σχολεία, έκλειναν κέντρα εργασίας και λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα. Τι θέλω να πω από αυτό. Ο ιός υπήρχε, ήταν κάτι καινούριο, ε, το είχαμε εντοπίσει ως ε, ένα καινούριο ιό ή τα έναν ή ένα, για τον οποίο δεν γνωρίζαμε κάτι και το μόνο που γνωρίζουμε ήταν ότι ήταν ιδιαίτερα μεταδοτικός και τους ε, πρώτους, τις πρώτες μέρες η θνησιμότητα ήταν στο 6% και δεν ξέραμε πώς θα συμπεριφερθεί. Ξέραμε όμως ότι έπλητε γρήπη ανθρώπους ε, υγιείς ενήλικες. Δηλαδή το 30% τουλάχιστον ήταν ε, υγιείς ενήλικες. Αυτό φυσικά έπρεπε να ανησυχήσει τις ε, αρχές ε, υγείας σε κάθε χώρα και από εκεί και πέρα ο το Επιδημιολογικό Κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μας είπαν ότι πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα και από εκεί και πέρα οι χώρες ε, βάσει του κανονισμού τους έπρεπε να προσαρμόσουν τα μέτρα αυτά στη χώρα τους. Εγώ ως υπουργό λοιπόν έπρεπε να λάβω όλα τα προληπτικά μέτρα προκειμένου να προλάβουμε την επιδημία και να μπορέσουμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της επιδημίας. Αυτή ήταν η ευθύνη μας και οι όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν μια προσπάθεια να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες και να χρησιμοποιήσουν και κοινά μέτρα για να μετριαστούν οι επιπτώσεις. Αυτό κάναμε και κάναμε κάτι καλό συναντηθήκαμε, οι Υπουργοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να συντονίσουμε κάποιες δράσεις. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι συμφωνήσαμε, για παράδειγμα, ε, για τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Κάτι το οποίο σήμερα το, έχουν, το θεωρούν όλοι δεδομένο, αλλά υπήρχε ε, συντονισμός μεταξύ των ε, αρχών, μεταξύ των Υπουργών Υγείας και των επιστημόνων για το ποιες είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου, ποια είναι, ε, ποιες ήταν οι ομάδες στις οποίες έπρεπε να εστιάσουμε πρώτα. Και ε, λάβαμε και κάποια μέτρα οργανωτικού χαρακτήρα. Το πιο διαφιλονικούμενο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι τα εμβόλια και κάθε χώρα έλαβε αποφάσεις ανάλογα με την ομάδα κινδύνου που ήθελε να προφυλάξει. Και όλες οι χώρες τελικά συμφωνήσαμε ότι θα εμβολιάσουμε τους ίδιους ανθρώπους, ε, τις ίδιες ομάδες υψηλού κινδύνου που εμβολιάζαμε και για την εποχιακή γρήπη. Συνήθως εμβολιαζόταν το 30% του πληθυσμού και επομένως λογικό ήταν για να προλάβουμε την νέα επιδημία να εμβολιάσουμε το ίδιο 30% του πληθυσμού για την ε, γρήπη τα 1 1. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι πρέπει να αναλυθεί αυτό που συνέβη και ξεκίνησε μια διαδικασία έρευνας. Εμείς περιμένουμε τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι ω αρχή υγείας ο στόχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ήταν να προειδοποιήσουν τα κράτη ώστε να λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό. Τώρα που ο δείκτης θνησιμότητας ε, είναι χαμηλότερος από το αναμενόμενο και η μετάδοση είναι χαμηλότερη από το αναμενόμενο, είναι πολύ εύκολο να κάνουμε αναλύσεις. Έχει τελειώσει η επιδημία και τουλάχιστον είμαστε σε θέση από άποψη επιστημονικών ενδείξεων να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για όλα όσα συνέβησαν. Και νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αφήσουμε τους επιστήμονες να εργαστούν και θα περιμένουμε και τους εμπειρογνώμονες να δούμε τι έχουν να μας πούν. Κάθε χώρα όμως νομίζω ότι οθέτησε τα μέτρα τα οποία θεωρούσε βάσει δεδομένων και των συνθήκων ότι ήταν και τα καταλληλότερα. Με ρωτήσατε και για τη χώρα μου. Στην περίπτωση της Ισπανίας, όπως έλεγε ο Πρόεδρος, δεν είχε σημασία το ότι ήταν η Ισπανία. Λίγο πολύ όλοι δράσαμε ανάλογα με την κατάσταση που είχαμε ενώπιόν μας. Σκεπτόμασταν πάντα την προστασία της υγείας των πολιτών μας. Και αυτό ήταν πάντα το πιο σημαντικό. Ε, και αν μας ρωτήσετε, υπήρχε, ήταν εύλογο να υπάρχει κατάσταση επιφυλακής. Ε, θυμηθείτε τις εικόνες που είχαμε εκείνες τις ημέρες, την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό, στην Αργεντινή. Θυμηθείτε τις εικόνες στην Ιαπωνία ή στην Κίνα. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να γίνει αυτή η προσπάθεια, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο τώρα που ίσως ε, η επιδημία δεν ήταν τόσο μεγάλη, να ήταν ακριβώς επειδή λήφθησαν και τα κατάλληλα μέτρα. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξηθούν οι δωρεές οργάνων. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, να χρησιμοποιήσουμε την κοινή μας εμπειρία και νομίζω ότι η Ευρώπη έχει ένα τεράστιο αποθεματικό εμπειρίας και έχουμε κάνει όλη τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για να αυξηθούν οι δωρεές. Κάτι επιπλέον σημαντικό, αυξήθηκαν οι δωρεές παρά το γεγονός ότι μειώθηκαν τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Ε, δόξα το Θεό να πούμε, μειώθηκαν τα ατυχήματα στους δρόμους, αλλά εμείς αυξήσαμε τις δωρεές, που σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί οι δωρεές μεταξύ ζώντων. Κάτι ακόμα το οποίο έχει ε, δώσει αποτελέσματα και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το λάβουμε υπόψη είναι η κατάρτιση των επιρογνωμόνων στην ενημέρωση ε, για, τις, ε, για τα άσχημα νέα ε, και το πώς επικοινωνούν με τους ασθενούς. Τα χρόνια έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η δωρεά οργάνων από ηλικιαμένα άτομα που εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ καλοί δωρητές. Έχουμε όμως εμπειρογνώμονες που ξέρουν πώς να διαβιβάσουν τα άσχημα νέα και πώς να ενημερώσουν για πολύ συγκεκριμένους ε, τομείς ε, του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα τους μετανάστες. Θα ήθελα να ξέρετε ότι στην Ισπανία υπάρχουν συγκεκριμένοι ε, μετανάστες, συγκεκριμένες ομάδες μεταναστών μπορεί να είναι από τους μεγαλύτερους δωρητές ε, στην Ισπανία παρά το γεγονός ότι στη χώρα τους δεν είναι δωρητές οργάνων. Λειτουργεί πολύ καλά το γεγονός ότι ε, δημοσιοποιούμε τα αποτελέσματα και οι πολίτες γνωρίζουν την ποιότητα, την ασφάλεια, την αλληλεγγύη και το γεγονός ότι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι ε, θα υπάρχει και κάποιο απόρριτο, θα, δεν, θα είναι εμπιστευτικέ οι πληροφορίες. Αυτό το φροντίζουμε καθημερινά. Τώρα, για τις συνέπειες των φαρμάκων. Υπάρχουν πολύ σημαντικά στοιχεία ε, για τα κατάλοιπα στα φάρμακα ε, η Ισπανία έχει ένα πρόγραμμα συλλογής πληροφοριών μέσω των φαρμακείων για τη διαχείριση και την ε, επεξεργασία αυτών των καταλήπων και τις συνέπειες που έχουν ε, στο περιβάλλον. Αυτό το πρόγραμμα ονομάζεται Σύγκρε και νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο θα μπορούσαμε να κάνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει το πολίτη είναι προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε τις πληροφορίες που μας λέτε για τους ε, υπαλλήλους της ΕΦΣΑ, ούτε για τη λειτουργικότητα της διατροφικής αλυσίδας. Ε, υπ' αυτή την έννοια ούτε στην Ισπανία, ούτε σε κάποιο άλλο κράτος μέλος μέσω του συστήματος ε, ε, διατροφικής επαγρύπνησης. Είναι κάτι το οποίο λειτουργεί καλά, το έχουμε όλοι στη χώρα μας και υπάρχει μια συγκεκριμένη ακρίβεια που μας προσφέρει μια ασφάλεια. Υπάρχει ένα σύστημα εκτάκτου ανάγκης ε, και από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει συγκεκριμένη διατροφική εκτακτή ανάγκη που αναφέρατε εσείς. Για τις εξαγωγές τροφίμων. Οι εξαγωγές πρέπει να τηρούν αυτό που ε, λένε οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Αυτό είναι θεμελιώδες για μας και αυτό περιλαμβάνουν και επιθεωρήσεις στην πηγή. Ε, κάποιο άλλο στοιχείο είναι οι περιβαλλοντικές ε, συνθήκες. Επιμένω όμως το κτηνιατρικό και διατροφικό, ο κτηνιατρικός και διατροφικός οργανισμός κάνει ελέγχους και επιτόπου και κάθε ε, χώρα κάνει και ελέγχους στα σύνορα. Ε, θα πρέπει ίσως να οργανώσουμε μία ημέρα για να συζητήσουμε τις εισαγωγές-εξαγωγές. Υπάρχει συγκεκριμένη ημέρα στη Σεβίλη ε, για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά, διότι πάντα υπάρχουν εκκρεμότητες. Και ολοκληρώνοντας, ε, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να πάρω ένα λεπτό για να απαντήσω κάποια θέματα τα οποία μου θέσατε για την οδηγία για τη διαμεθοριακή περίθαλψη να διευκρινίσω κάτι που ίσως όλοι εσείς γνωρίζετε. Ο κανονισμός 883 του 2004 και που θα τεθεί σε ισχύ φέτος το 2010. Αυτή τη στιγμή εγκριθούν οι εφαρμοστικοί κανονισμοί 987-989 του 2009 θα απαντήσουν σε πάρα πολλά θέματα τα οποία έθεσε η νομολογία. Δεν λέω από τις ανάγκες των πολιτών, αλλά ε, που θα μπορούσαν να θέτουν και μέσω ε, ημών, αλλά από κάποια πράγματα που έχουν προκύψει από την ομολογία. Λίστε αναμονή. Κανονισμό ε, σημείο 2 του 883 λέει ότι υπάρχει δικαίωμα περίθαλψη εάν περιλαμβάνεται μεταξύ των θεραπείων τη χώρα διαμονή και δεν και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση από ιατρικής πλευράς. Αυτό περιλαμβάνεται στον κανονισμό. Δεύτερον, οι χρονικές συγκυρίες σε άλλη χώρα, ε, ε, αυτή της χώρας ε, διαμονή. υπάρχει το δικαίωμα της κάρτας ασθενούς και υπάρχει δικαίωμα περίθαλψης. Αυτό το λέει το άρθρο 19 του 883. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ετοιμάσει και τον κατάλογο των ε, παροχών υγείας ε, που είναι τελείως ε, διαφορετικός από αυτόν που έχουμε. Επίσης, στο άρθρο 16 του 883 λέει ότι η ρήθαλψη θα γίνεται βάσει του κανονισμού της χώρας διαμονής. Και υπάρχει και η πρώτερη έγκριση από πλευράς της αρμόδιας αρχής. Αυτό στην οδηγία για τους ασθενείς. Επομένως, η περίθαλψη και η κινητικότητα βάσει αυτών που μας ζητά το δικαστήριο ρυθμίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν εκτόσεις που καθορίζουν αυτή τη συγκεκριμένη απέτηση για πρώτερη έγκριση. Να σας πω όμως το εξής. Εγώ θέλω να έχουμε μία διαμεθοριακή οδηγία για την περίθαλψη. Σας είπα στην αρχή που θε, ότι θέλουμε μία οδηγία που θα είναι φιλόδοξη, που θα ρυθμίζει ένα πακέτο περίθαλψης, το οποίο θα είναι κοινό για όλες τις χώρες, γιατί θα σας πω το εξή. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι η οδηγία, όπως μας παρουσιάστηκε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν έδινε ενιαία και ομογενή περίθαλψη σε όλους τους πολίτες. Όχι. Όταν ένας ασθενής από τη μία χώρα πήγαινε σε άλλη χώρα για να λάβει κάποια θεραπεία, του καλύπτονταν μόνο ε, τα έξοδα για την περίθαλψη που μπορεί να λάβει και στη χώρα του. Μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά δεν καλύπτονταν όλες οι παροχές υγείας, αλλά μόνο ό,τι μπορούσε να λάβει και στη χώρα του. Που σημαίνει ότι η αποζημίωση θα δινόταν μόνο σε σχέση με αυτό που ελάμβανε στη χώρα του. Δεν περιλαμβάνε, ε, ένα πακέτο το οποίο ήταν προς το κοινό συμφέρον των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Για παράδειγμα, αποκλειόνταν ε, ε σπάνιες ασθένειες για τις οποίες χρειάζονται συγκεκριμένα νοσοκομεία ευρωπαϊκά για τη θεραπεία τους. Δεν χρειαζόταν πρώτερη έγκριση του ιατρού για έναν ασθενή. Ένας ασθενής μπορούσε να επιλάξει χωρίς καμία ε, ιατρική συμβουλή και να πάει σε μια χώρα να λάβει περίθαλψη χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο και για, σε, ποιο, ε, σε ποια χώρα. Γιατί δεν υπήρχε έλεγχος ποιότητας και διασφάλισης σε ένα νοσοκομείο, σε ένα κέντρο το οποίο να βρισκόταν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Υπάρχει ανάγκη λοιπόν ποιότητας εναρμόνισης των υπηρεσιών υγείας και στόχος είναι να το συμπεριλάβουμε αυτό στο επόμενο Συμβούλιο όταν θα συζητηθεί το θέμα και μαζί με τις υπόλοιπες χώρες μέλη. Πρόκειται για θέματα τα οποία πάνε λίγο παραπέρα, διότι πρέπει να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε την ιατρική περίθαλψη. Να έχουμε ένα πακέτο υγείας που θα διασφαλίζει κάποιες ελάχιστες υπηρεσίες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Frau Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για όλες τις απαντήσεις. Έχουμε μπροστά μας πολλές ζωντανές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. θα πρέπει σιγά σιγά να διευκρινίσουμε για τι πράγμα μιλάμε, να περάσουμε σε μεγάλα θέματα, εναρμόνιση υγειονομικών υπηρεσιών παραδείγματο χάρη. Ξέρουμε ότι είναι Ηράκλειος άθλος το να συζητάμε τέτοια θέματα στις 27 χώρες μέλη. Μας είπατε ότι θα είστε μία ειλικρινής ε, μεσάζων σε αυτά τα θέματα και χαιρόμαστε που θα ασχοληθείτε με αυτό το θέμα. Ξέρουμε ότι εκατομμύρια πολιτών ζητούν ε, να καταλάβουν την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα θέματα της υγείας. Είναι κρίμα να υπάρχουν σύνορα, να υπάρχουν υπαλλήλοι φραγμοί στον τομέα της υγείας. Θα έχουμε το χρόνο όμως να ξανασυζητήσουμε τα θέματα αυτά σε πολλές ευκαιρίες. Ξέρω ότι ε, έχετε συζητήσει το θέμα αυτό ε, και με τους συντονιστές ε, και έχετε κάνει και συναντήσεις προετοιμασίας. Ξέρω ότι είστε ενθουσιώδεις για τον τομέα σας και περιμένουμε, προσβλέπουμε στις μελλοντικέ συζητήσεις μας. Είναι πολλά θέματα τα οποία είναι και για σας σημαντικά και για μας σημαντικά. Καλή σας επιτυχία λοιπόν και θα σας ξαναδούμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ευχαριστούμε για την επισκεψή σας. Okay, goodbye. Okay. Wir kommen zum nächsten Punkt der Και εμείς περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το υπαριθμό 19, και μένουμε στο θέμα που ήδη αρχίσαμε να συζητάμε. Πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση. Έχουμε έναν εισηγητή που έχει ασχοληθεί εις βάθος με αυτό το θέμα, ο μιροσλάβ Μικολάσιτς, στον οποίο θα δώσω κατευθείαν το λόγο. Ας περιμένουμε μισό λεπτάκι για να ησυχάσει η αίθουσα. Ja, das war alles sehr interessant und aufregend, aber die Gespräche... Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αλλά τώρα οι περαιτέρω συνομιλίε θα γίνουν εκτό αιθούση για να μπορέσουμε και εμεί να συνεχίσουμε. Okay, ich glaube, jetzt können wir okay. weitermachen. Bitte. Uh, Mr. President, dear colleagues. Um, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να επωφεληθώ τη ευκαιρία ε, για να μιλήσω για την πρόταση τη Επιτροπή, που είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών εργασιών και δημοσίων διαβουλεύσεων. Όπω είδαμε κατά την δημόσια ακρόαση για την ασφάλεια και την ποιότητα των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση το Νοέμβριο του 2009, αυτή η πρόταση ε, είναι μια πρόταση που μπορούμε να χαιρετήσουμε και εμεί και όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Να πω δύο λόγια για την πρόταση αυτή καθεαυτή πριν μιλήσω για κάποιες ιδιαιτερότητες και για τις τροπολογίες που προτείνω στην έκθεσή μου. Η προτινόμενη οδηγία θέτει κανόνες για να διασφαλίσει υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας για όργανα που προορίζονται για μεταμόσχευση. Και μιλάμε για τις διαδικασίες δωρεάς, ε, αφαίρεση ελέγχου χαρακτηρισμού συντήρησης μεταφοράς και μεταμόσχευσης. Η οδηγία εισάγει εθνικά προγράμματα ποιότητα που προσδιορίζουν κανόνε και πρακτικέ για τη διαδικασία μεταμόσχευση στα κράτη-μέλη και αναλύει λεπτομερέστερα τη διαδικασία απόκτηση και τα όσα αφορούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και προβλέπει ένα σύστημα υποβολή στοιχείων. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανιχνευσιμότητα και την προστασία του δότη και του λήπτη. Όσον αφορά την εφαρμογή, υπάρχουν διατάξει σχετικά με τον ορισμό και τα καθήκοντα των αρμοδίων εθνικών αρχών, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ανταλλαγή Οργάνων και την ανταλλαγή οργάνων με τρίτε χώρε. Για να διασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασία τη υγεία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η προτινόμενη οδηγία καθορίζει κοινά δεσμευτικά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση. Και μετά την έγκριση της οδηγίας για την ποιότητα και ασφάλεια αίματος ε, και προϊόντων αίματος το 2003, μετά την οδηγία για την ποιότητα και ασφάλεια ανθρωπίνων ιστών το 2004 και κυτάρων, αυτή η οδηγία προσπαθεί να συμπεριλάβει και τα ανθρώπινα όργανα για να ολοκληρώσει την οδηγία με βάση το άρθρο 168 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Χρειάζεται κοινή δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίστηκε σαφώς στο ψήφισμα για την μεταμόσχευση και τις δωρεές που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία τον Απρίλιο του 2008. Η μεταμόσχευση οργάνων ε, τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει ε, μια πρακτική παγκοσμίως αποδεκτή που βελτιώνει την ποιότητα ζωής και επεκτείνει το προσδόκιμο ζωής. Η δωρεά ε, οργάνων είναι έκφραση αλτρουισμού και αλληλεγγύης στην κοινωνία. Παρ' αυτά, η ανάγκη για μεταμόσχευση οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι σταθερά αυξάνεται πιο γρήγορα από τον αριθμό οργάνων που είναι αντικείμενο δωρεάς. Σημαντικός αριθμός ασθενών ε, αποβιώνουν λόγω της χρόνιας έλλειψης οργάνων. Έχουμε έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των αναγκών και της διαθεσιμότητας οργάνων που μπορεί να οδηγήσει σε εμπορευματοποίηση και παράνομη διακίνηση οργάνων, πράγμα που παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η έλλειψη οργάνων παραμένει η πιο σημαντική πρόκληση και υπάρχουν ε, πολλές ε, λεπτομέρειες ανάλογα με τα διάφορα συστήματα μεταμόσχευσης που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη-μέλη. Η ενισχυμένη συνεργασία και οι διασυνοριακέ ανταλλαγέ μεταξύ κρατών μελών παρουσιάζουν σημαντικό δυναμικό για την αύξηση του αριθμού των μεταμοσχεύσεων και αυτό απαιτεί την έγκριση κοινών προτύπων ποιότητα και ασφάλεια. Χαιρετίζω λοιπόν την πρόταση αυτή και θεωρώ ότι είναι σημαντική οι τρεις βασικοί στόχοι. Διασφάλιση τη ποιότητα και ασφάλεια για του ασθενεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφάλιση προστασία των δωρητών και διευκόλυνση τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει συνένεση για την δωρεά οργάνων, για το σκοπό της μεταμόσχευσης. Ωστόσο, λόγω των διαφορετικών πολιτιστικών ε, συστημάτων και τη διαφορετική οργάνωση, υπάρχουν διαφορέ μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την προσέγγιση στα θέματα αυτά προσπαθούμε να κινηθούμε προς την εναρμόνιση των μέτρων ποιότητας και ασφάλειας, αλλά παρόλα αυτά τονίζω ότι η οδηγία δεν πρέπει να δημιουργεί ένα επιπλέον διοικητικό άχθος για τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να παραμείνει η ευελιξία χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι τωρινές καλές πρακτικές. Θέλω να τονίσω κάποια σημαντικά θέματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις προτινόμενες τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσής μου. Καταρχήν, κοινός μας στόχος είναι τα κοινά πρότυπα για την ποιότητα και την ασφάλεια οργάνων για μεταμόσχευση. Κοινά πρότυπα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύτερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη που ήδη έχουν καλά συστήματα υγείας και μεταμοσχεύσεων θα πρέπει να μπορούν να διατηρήσουν τις οργανωτικές και διοικητικές τους δομές. Παράλληλα, η οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν ή να εισάγουν πιο αυστηρά προστατευτικά μέτρα από αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν. θα τηρούμε ε, το είδος της οργάνωσης, ε, θα σεβόμεθα το είδος οργάνωσης που έχουν ε, τα κράτη-μέλη και θα αποφεύγονται παρεμβάσει τη κοινότητα σε τομεί εθνική κυριαρχία. Θα κρατήσουμε αυτά τα οποία ήδη λειτουργούν σωστά στην πράξη. Δεύτερον, όσον αφορά την ασφάλεια, της δωρεάς οργάνων και της μεταμόσχευσης, η έννοια της ανωνυμίας θα πρέπει να αντικατασταθεί από την έννοια της ανιχνευσιμότητας. Δηλαδή κάθε όργανο θα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμο από το δότη προς το λήπτη και αντιστρόφος Η έννοια της ανιχνευσιμότητας και της δυνατότητας ταυτοποίησης συνδέονται στενά και όταν μιλάμε για την ανιχνευσιμότητα του κατόχου του βιολογικού υλικού, αυτός ο κάτοχος του βιολογικού υλικού θα πρέπει να μπορεί να ταυτοποιηθεί και σε αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δότες και οι λύτες. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ε, την εμπιστευτικότητα και την ακαιρεότητα ε, ε, καθώς και τη διαθεσιμότητα προσωπικών δεδομένων δοτών και λιπτών. Τρίτο σημείο οικειοθελής ε, και ανιδιοτελής δωρεά οργάνων, χωρίς αμοιβή. Συμφωνώ με την ε, άποψη της Επιτροπής ότι τα, τα προγράμματα μεταμόσχευσης οργάνων βασίζονται στην αρχή της οικειοθελούς ε, δωρεάς χωρίς αμοιβή. Αυτή η έννοια ήδη υπάρχει στην μέχρι τώρα νομοθεσία για τις ουσίες ανθρώπινης προέλευσης η δωρεά οργάνων θα πρέπει πάντοτε να είναι χωρί αμοιβή και να μην υπάρχει καμία σύνδεση με πιθανή εμπορευματοποίηση. Επιπλέον, η δωρεά και τα συστήματα μεταμόσχευση βασίζονται στον αλτρουισμό. Υπάρχει σχέση μεταξύ της αρχής τη οικειοθελού ανιδιοτελού δωρεά και τη ποιότητα και ασφάλεια ε, από την άλλη πλευρά. Όταν η δωρεά δεν είναι οικειοθελή και προβλέπεται και κάποιο οικονομικό όφελο, η ποιότητα τη διαδικασία δωρεά δεν μπορεί να είναι πλήρω εγγυημένη εφόσον η βελτίωση της ποιότητας ζωής ή ε, η ε, διάσωση της ζωής ενός ατόμου δεν είναι ο κύριος στόχος ή ο μοναδικός στόχος που θέλουμε να επιτευχθεί σχέση μεταξύ της παραβίασης ε, των αρχών της οικειοθελούς και μη εμπορευματοποιημένη δωρεάς οργάνων δίδεται από την περιγραφή των της έκβασης των μεταμοσιεύσεων όταν έχουμε πράξεις εμπορευματοποίησης ε, και εμπορίας οργάνων ή εμπορίας ανθρώπων με στόχο την αφαίρεση οργάνων. Εδώ έχουμε ένα μοντέλο τέτοιας παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών αρχών ηθικής και διοντολογίας που θα έπρεπε να διέπουν τις ε, δωρεές οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις όπως αναφέρεται και από τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ιατρικής και το πρόσθετο πρωτόκολλο για τους ιστούς ανθρώπινης προέλευσης. Όπως επίσης και στις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΗ για τις μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων οργάνων. Αυτή η αρχή δηλώνεται και ε, στο Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συμπεριλήφθηκε και στην οδηγία του 2004 23 του 2004 για ιστούς και κύτταρα και την οδηγία 98 του 2002 για το αίμα και, και προϊόντα αίματος. Και οι τρεις οδηγίες βασίζονται στο ίδιο άρθρο, το 168 της συνθήκης και πολλοί δωρητές οργάνων είναι και δωρητές ιστών. Επομένως, ε, θα ήταν παράλογο να μην διατηρήσουμε την ίδια αρχή και στην τωρινή μας νομοθεσία. Ε, θα ολοκληρώσω την παρέμβασή μου, πρώτα, δεν θα αργήσω. Τέταρτο σημείο. Όσον αφορά την προστασία του δότη και του λήπτη, προτείνω κάποιες τροπολογίες ε, για τη σχέση μεταξύ δοτών εν ζωή και μεταθανάτιων δοτών, για να έχουμε καλύτερη ποιότητα και ασφάλεια. Στόχος είναι η διασφάλιση του ότι ο δυνητικός εν ζωή δότης θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να κάνει ε, μια ελεύθερη επιλογή σχετικά με την ε, δωρεάν χωρίς να υπάρχουν ιατρικές, ψυχολογικές ή κοινωνικές επιπλοκές σε σχέση με τη δωρεά και στη συνέχεια να εξασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη φροντίδα για τον δότη και η μη επακολούθηση επιπλοκών από την δωρεά οργάνων. Η οποιαδήποτε αντιστάθμιση θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην κάλυψη δαπανών όπως ε, δαπάνες ε, ταξιδίου ή απώλεια εσόδων, αλλά να μην συμπεριλαμβάνονται καθόλου οικονομικά κίνητρα για τη δωρεά οργάνων. Ε, και κάποιος ο οποίος έχει υποστεί αδικαιολόγητη βλάβη λόγω της δωρεάς οργάνων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποζημίωσης ε, που πάλι θα περιορίζεται αυστηρά στην αντιστάθμιση της ζημίας που υπέστη από τη δωρεά οργάνου. Εδώ θέλω να τονίσω ότι δεν τίθεται σε αμφισβήτηση η αρχή της οικειοθελούς και ανιδιοτελούς δωρεάς. Αυτό εντάσσεται στο άρθρο 15, προστασία του ενζοηδότου. Και πέμπτον, τελευταίο σημείο, για να βελτιώσουμε τη διαδικασία μεταμόσχευσης, προτείνω πιο συγκεκριμένη διατύπωση σε κάποια άρθρα για να βελτιώσουμε το κείμενο. Αυτά όσον αφορά τον ορισμό του δότη, της αρμόδιας αρχής, της περίοδου μετά τη μεταμόσχευση και κάποιες άλλες έννοιες. Κλείνω κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι και θέλω να σας πω ότι πιστεύω ότι οι κοινέ ε, βέλτιστες πρακτικές ε, και τα μοντέλα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρήσιμα για την αύξηση του αριθμού των δωρητών. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία, ούτως ώστε να εντοπίσουμε τις επιτυχίες των συστημάτων μεταμόσχευσης και να τις προωθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα μας οδηγήσει σε, βελτιωμένη, σε ένα βελτιωμένο σύστημα στην παροχή οργάνων δωρεάς Ευχαριστώ για την προσοχή σας αγαπητοί συνάδελφοι και με σίγουρος ότι θα έχουμε πολλές επικοδομητικές συζητήσεις και θα περιμένω τα σχόλιά σας και τις προτάσεις σας για την πρόταση της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μικολάσιτ, λέει ο Πρόεδρος. Καλή επιτυχία για την έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ που ασχοληθήκατε εντατικά και αποτελεσματικά με αυτό το θέμα. Φαίνεται ότι το θέμα αυτό ε, υπό την τρέχουσα προεδρία θα καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχουμε τους ομιλητές. Ανδρέας Περέγιο, πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η οδηγία που μας παρουσίασε με την έκθεσή του ο κύριος Μικολάσιτς είναι μια οδηγία την οποία θεωρούμε απαραίτητη και μια καλή βάση. Θα ήθελα να αναγνωρίσω δημοσίως το έργο του εισηγητή και την στάση την οποία κράτησε κατά τη διάρκεια των εργασιών, γιατί μπορέσαμε να έχουμε έναν επικοδομητικό διάλογο, καρπός του οποίου φαίνεται και από την ακρόαση που κάναμε, που μας έδωσε τη δυνατότητα για συζήτηση, υπήρχε ανα πάσα στιγμή καλός συντονισμός, ε, και ε, ως εισηγητής ε, και με την έναρξη της Ισπανικής Προεδρίας για να δούμε τι γίνεται και πόσο καλή δουλειά έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι λόγοι ε, για αυτή την οδηγία, για τις λίστες αναμονής που έχουμε ε, για τη μεταμόστευση οργάνων, τις ε, ποσότητες των οργάνων που έχουμε για δωρεά στις διάφορες χώρες, το γεγονός ότι η έλλειψη οργάνων δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, πρέπει να κάνουμε κάτι και όλα αυτά τα θέτουμε γνωρίζοντας ε, στα πλαίσια των ετών και ποια είναι τα αποτελέσματα των ε, δωρεών. σώζονται ζωές, ε, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής κάποιου και ε, να ξέρουμε και ότι με, τα, με όλες οι μεταμοσχεύσεις, λαμβάνοντας για παράδειγμα τη μεταμόσχευση νεφρών, έχουν μια σχέση κόστους ποιότητας η οποία είναι εξαιρετική. Συμφωνώ λοιπόν με όσα είπε ο κύριος Μικολάσιτς και είναι σαφές ότι η οδηγία πρέπει να αναζητήσει και προσπαθεί να εξεύρει έναν τρόπο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, να βρει καλύτερα όργανα, να βελτιώσει την ποιότητά τους και να έχουμε και ένα ευρωπαϊκό αν θέλετε σύστημα το οποίο θα είναι πιο προσβάσιμο, πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό. Υπάρχουν βέβαια κάποιες πτυχές τις οποίες θα πρέπει να φροντίσουμε ιδιαίτερως. Ε, καταρχάς ε, έχουμε λίγο περιορισμένο χρόνο και για να μπορέσουμε να καταθέσουμε τροπολογίε, θα πρέπει να κάνουμε πολύ καλή δουλειά για να μπορέσουμε να έχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Ε, τα άρθρα 13 και 15 θα ήθελα να αναφέρω, ε, στα οποία περιλαμβάνονται πτυχές που αφορούν την ε, δωρεάν ε, δωρεά οργάνων, το να γίνεται θελουσία βάση, και να υπάρχει μια σαφής διαδικασία δωρεάς και κυρίως ε, το τι γίνεται με τη δωρεά εν ζωή. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ περισσότερο, διότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες απόψεις ε, ε, που να ερίζουν στο θέμα αυτό. Μπορεί να είναι μια δωρεά συμπληρωματική της δωρεάς που γίνεται μετά θάνατον, αλλά ε, σίγουρα θα είναι και η ίστατη λύση εάν δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ε, δωρεάς μεταθάνατων. Θα πρέπει λοιπόν να τα φροντίσουμε ιδιαίτερως να μην υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ της οδηγίας και των εθνικών ε, προγραμμάτων δράσης που θα συζητήσουμε αργότερα. Εγώ προσωπικά να σας πω ότι στα πλαίσια της συνεργασίας θα ήθελα να παρουσιάσω κάποιες τροπολογίες επί του θέματος. Όσον αφορά τώρα την ποιότητα των ε, οργάνων, είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να έχουμε μόνο το θέμα της προστασίας δεδομένων αποκλειστικά. Ναι, μεν είναι αλήθεια ότι πρέπει να προστατεύονται τα δεδομένα, αλλά επίσης από ιατρικής πλευράς χρειάζεται και αυτό που είπε ο κύριος ε, ε, Μικολάσιτς να έχουμε τη δυνατότητα ανιχνωσιμότητας των οργάνων και ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να παραμείνουν ιατρικό απόρριτο ακριβώς γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ποιότητα του οργάνου και πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι ο ασθενής, τι ασθένειες μπορεί να είχε και τι ακριβώς ε, προέκυψε και από την επίδραση φαρμάκων. Όλες αυτές οι πληροφορίες ναι μεν είναι ε, απόρριτες από ιατρικής πλευράς αλλά πρέπει να τις γνωρίζουμε για την ποιότητα των οργάνων. Υπάρχουν δυνατότητες λοιπόν για μεγάλες ελλείψεις και είναι κρίμα ε, η τόση πολύ καλή δουλειά που έγινε μέχρι τούδε να πάει χαμένη. Γι' αυτό ελπίζουμε να οδηγηθεί σε αίσιο τέλος και να εγκριθεί αυτή η οδηγία σε πρώτη ανάγνωση. Υπάρχει διάθεση για διάλογο, δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ ημών και ημών και ε, η οδηγία είναι καθόλου επίκαιρη παρά το γεγονός ότι πάντα ε, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και εγώ πιστεύω ότι και τα εκτιμώντας θα μπορούσαμε να τα διευρύνουμε λίγο διότι στα εκτιμώντας ε, καθορίζεται ποιος είναι ο στόχος μας. Ίσως όμως θα έπρεπε στα εκτιμώντας να περιλαμβάνονται και κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες και να εξηγούν λίγο καλύτερα τι ακριβώς έχουμε στο διατακτικό του κειμένου, διότι χρειαζόμαστε παιδεία στο θέμα των μετανοσχεύσεων, όχι μόνο στις χώρες μέλη που θα αναλάβουν το θέμα του συντονισμού, αλλά και για τους επαγγελματίες οι οποίοι θα δρούν επί του θέματος και φυσικά και οι πολίτες που πρέπει να γνωρίζουν την οδηγία. Δεν θα πρέπει λοιπόν να λησμονούμε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το ε, χέρι μας για να έχει και κάποιο εκπαιδευτικό ρόλο αυτή η οδηγία. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Να συγχαρώ για άλλη μια φορά τον εισηγητή για τη δουλειά του και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την αγαστή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιανακουδάκη. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για αυτή την έκθεση που είναι πλήρης και πολύ ευαίσθητη για αυτό το θέμα που είναι πολύ δύσκολο ε, για πολλούς λόγους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο αριθμό δωρητών είναι σχετικά χαμηλός σε σχέση με τη ζήτηση που υπάρχει. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μιλάμε για 28% ε, κάλυψη και κατά μέσο όρο πεθαίνουν τρία άτομα κάθε εβδομάδα εν αναμονή μεταμόσχευσης. Η κατάσταση ποικίλει σε κάθε κρατό μέλο ανάλογα ε, με τι υπηρεσίε που προσφέρονται και αυτή η έκθεση προσπαθεί να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα προτείνοντας ομοιόμορφες ε, διατάξεις για πολλά κράτη-μέλη, κάποια σταθερά πρότυπα τα οποία θα βελτιώσουν ε, την ποιότητα και ελπίζουμε ότι θα αυξήσει τον αριθμό των ε, δωρητών. Και επίση ένα στόχο είναι η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη όλων στον τομέα. Με χαροποιούν φράσεις ε, ε, όπως την τροπολογία 11 που λέει ότι δωρητής μπορεί να είναι είτε εν ζωή είτε μεταθανάτιος. Το ανθρώπινο σώμα είναι το σώμα ενός ε, ατόμου ακόμη και μετά θάνατον. Υπάρχουν ενδιαφέροντα σημεία, η αναγνώριση και η προσέγγιση στην προστασία των δεδομένων. Νομίζω ότι παρουσιάζει μια καλή ισορροπία και ενδυναμώνει την οδηγία. Οι τροπολογίες για τα όργανα για χώρες του τρίτου κόσμου επίσης είναι σημαντικές. Θέλουμε να έχουμε μια ισχυρή οδηγία για την εμπορία των οργάνων. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί και από το σχέδιο δράσης το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και νομίζω ότι μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο μας. Συγχαίρω λοιπόν άλλη μια φορά τον εισηγητή και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει ομόφωνα αυτή την έκθεση. Ευχαριστούμε κυρία Ματίας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή για τη δουλειά του και να τον συγχαρώ. Νομίζω το θέμα είναι άκρο σημαντικό, όπως αναφέρθηκε επανειλημμένος. Είναι πολλά τα ζητήματα στα οποία συμφωνούμε, οπότε δεν θα σταθώ σε αυτά. Νομίζω ότι η δουλειά που κάνατε ήταν πολύ αυστηρή, πολύ μεθοδική και πραγματικά σας συγχαίρω ξανά. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα για το οποίο παραμένουν κάποιοι από τους μου. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε το ζήτημα αυτό κατά μέρος, θα πρέπει να εμβαθύνουμε κι άλλο και έχει να κάνει με την αντικατάσταση που προτείνεται της ανωνυμίας με αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας. Θεωρώ ότι για να διασφαλίσουμε την προστασία των πολιτών, κάτι που είναι για μας καθοριστικό, και για να βάλουμε στον υψηλότερο δυνατό επίπεδο την ποιότητα που θα επιδιώκουμε, για, τα, για τους λήπτες ε, των οργάνων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη μεταμόσχευση, Νομίζουμε ότι εδώ πρέπει να διασφαλίσουμε οπωσδήποτε την ανωνυμία. Αυτό το βρίσκουμε θεμελιώδου σημασία. Και στο επίπεδο του δότη και γενικώ. Και ελπίζουμε ότι η Επιτροπή θα το λάβει αυτό υπόψη και θα καταφέρει να ευθυγραμμίσει τι απαιτήσει τη ανωνυμία με την εμπιστευτικότητα. Δεν ξέρω αν είναι συμβατά τα μέτρα που προτείνονται τώρα, αλλά ελπίζω ότι θα γίνει η συζήτηση ώστε να εμβαθύνουμε και να δούμε που υπάρχει ασυμβατότητα εφόσον κάτι τέτοιο ισχύει και πώς θα μπορέσουμε να τις καταπολεμήσουμε. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αμφισβητήσουμε εδώ την ελάχιστη εγγύηση ότι τα συστήματα να είναι στο δυνατόν πιο διαφανή και να μην περιορίσουμε τη δυνατότητα ανοίγματο του συστήματο στη σωστή κατεύθυνση όμω Να μην επιτρέψουμε να παρισφύσουν προβλήματα τα οποία δεν θέλουμε να δούμε, να προκύπτουν. Να έχουμε λοιπόν ένα σύστημα πιο αυστηρό αλλά και πιο εύχριστο. Να χρησιμοποιηθεί λοιπόν η αρχή της ανωνυμίας. Για μένα είναι θεμελιώδης και βασική. Για τα υπόλοιπα ζητήματα νομίζω ότι εύκολα θα τα, θα τα συζητήσουμε και σε άλλες ευκαιρίες και θα καταλήξουμε και σε συμφωνία. Ευχαριστώ. Das waren Δώσαμε το λόγο στους ηγητές. Έχω και εγώ μια ερώτηση στην τροπολογία 27. Σωστά, κύριε Μικολάσιτς, ε, μιλάτε για τα συστήματα των κρατών μελών Ε, σχετικά με την καταγραφή των πιθανών δωρητών. Και οι αρμόδιες αρχές ε, δίνουν προτεραιότητα στις επιθυμίες ε, του δωρητού. Στα αγγλικά λέει competent authorities Και αυτό που λέγεται στα γερμανικά ακούγεται σαν, κρατικές, σαν κρατική αρχή, ενώ στη Γερμανία και σε άλλες χώρες είναι φορείς που είναι οργανωμένοι σε ιδιωτικό επίπεδο. Είναι αρχές δημοσίου ελέγχου, αλλά δεν είναι κρατικές αρχές, είναι ιδιωτικοί φορείς. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε τη διατύπωση που θα χρησιμοποιήσουμε. Να πούμε αρμόδιες αρχές και οργανισμοί, πάντως κάτι το οποίο στην γερμανική μετάφραση τουλάχιστον να εκφράζει αυτό το οποίο ισχύει και στη χώρα μου και σε άλλες χώρες. κυρία Αντώνια Παρβανόβα. Thank you, Mr. President. Uh, actually, uh, Ευχαριστώ, πρόβλημα. Εδώ, πρόεδρε, εδώ ο σχέδιος είναι η κυρία Φεδρική, η οποία μου ζήτησε να παρουσιάσω τις απόψεις της και να σχολιάσω εκ μέρους της την έκθεση του κυρίου Νικολάσικ. Έτσι λοιπόν εκ μέρους της θα συγχαρώ τον κύριο Νικολάσιτ, διότι το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και περίπλοκο. Είναι τεχνικό το ζήτημα. Και είναι δύσκολο να εξεύρει κανεί την σωστή ισορροπία μεταξύ τη δημόσια ε, ζήτηση και των ιατρικών μεριμνών. Όμω, εκτιμούμε ιδιαίτερω το σχέδιο έκθεση που ετοίμασε ο κ. Μικολάσιτ. Είναι μια καλή βάση εργασία και ω και ο ε, τη ΑΛΔΕ ε, ε, συμφωνούμε με την απόφαση του να εμπλέξει όλε τι πολιτικέ ομάδε ήδη σε αυτή τη φάση τη συζήτηση. Ο κ. Μικολάσιτ θέλει οδηγία να είναι στο δυνατόν πιο ευέλικτη και οι επαγγελματίες του τομέα υγείας να έχουν την τελική απόφαση για τις ανάγκες και τα κριτήρια που θα ταυτοριστούν. Το σχέδιο έκθεσης καλεί την ευρύ φάσμα σημαντικών ζητημάτων και για την ομάδα ΑΛΔΕ, όπως η ευελιξία, το πεδίο της οδηγίας, ο ρόλος των ειδικών αρχών, και η ενισχυμένη τους συνεργασία, ο πλήρης σεβασμός τριών αρχών, της ομοφωνίας, της ανταμοιβή των ζώντων δοτών και τη στήριξη των θανάτων δοτών. Εδώ είμαστε όμω σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή που ασχολείται με ζητήματα υγεία και θέλει να βελτιώσει τα δικαιώματα των ασθενών. Λόγω τη βιοτεχνολογία και των καλύτερων δυνατών διατηθέμενων ιατρικών πρακτικών, κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Επίση, θα πρέπει συγκεκριμένα να αναφερθεί η έκκλησή μα για την ε, κάρτα των Ευρωπαίων δοτών που να συμπληρώνει τα εθνικά συστήματα. Τώρα, σε λεπτομέρειε για τα βασικά ζητήματα, να αναφέρω απλώ ότι θέλουμε να ληφθεί υπόψη η μεταφορά ω νέα, νέα ιατρική ειδικότητα που θα πρέπει να χρησιμοποιεί τι καλύτερε δυνατέ γνώσει και τι πλέον προηγμένε ιατρικέ τεχνολογίε ώστε να διασφαλίζουμε όλου ε, του κινδύνου και τι απειλέ που μπορεί να προκύψουν από τη μεταφορά του οργάνου, ε, ιδίω στην ε, αποβολή. Και τι τροπολογίε 1 και 5 να ξαναδούμε. Επίση, οι οργανώσει ε, ασθενών και όπω αναφέρεται και στο άρθρο 22 είναι σημεία που μα προκαλούν το εξή σχόλιο. Πρέπει να διερευνήσουμε πόσο η οδηγία θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να διατηρήσουν τι υπάρχουσε σχέσει του με του ευρωπαϊκού οργανισμού ανταλλαγή οργάνων όπω η Eurotransplant και θα προτείνω μια τροπολογία για το άρθρο 22 προκειμένου να διευκρινίσουμε τι δυνατότητε και το πεδίο αυτή τη συνεργασία. Για το πεδίο τώρα συγκεκριμένα τη οδηγία, στηρίζουμε την ιδέα του κυρίου Μικολάσιτ, το πεδίο να παραμείνει στη διασυνοριακή μεταφορά των οργάνων στις τροπολογίες 5 και 41 και τον στηρίζουμε και στην ιδέα να προσθεθεί η περίπτωση της αποβολής οργάνων ή της ανάγκης περίθαλψης. Τώρα για την μη αμοιβόμενη δωρεά, στο άρθρο 14 της ε, οδηγίας ορίζεται ότι η δωρεά από ζώντες δότες θα πρέπει να γίνεται και ο θελός βεβαίως και στις 22 Απριλίου 2008 υπάρχει και μια έκθεση που δημοσιεύτηκε σχετικά, η έκθεση Άνταμο, όπου ορίζονται οι, οι προποθέσει υπό τι οποίε τα κάτι μέλη μπορούν να προβλέψουν και αμοιβέ για τη δωρεά οργάνων. Εδώ μιλάμε για ιατρικές και κοινωνικέ ανταμοιβέ, όχι πληρωμή για τους δωρητές. Η ομάδα Άλντε λοιπόν για το σημείο αυτό έχει δύο αιτήσει. Πρώτα απ' όλα, να παραμείνουμε στη συμβαστική λύση που πετύχαμε στην απόφαση του 2008 στην παράγραφο της 22 και ακριβώς γι' αυτό προτιμούμε τη διατύπωση που, προτείνει ο κ. Περάγιο για την παράγραφο... στην παράγραφο 12 της δικής του... δικού του σχεδίου έκθεσης. Θέλουμε επίσης να συμπτύξουμε τις τροπολογίες 25 και 32 γιατί αφορούν το ίδιο ζήτημα και να ζητήσουμε όχι μόνο να υπάρχει ανταμοιβή, αλλά και πραγματική απολαβή για του ζώντε δότε. Εδώ τονίζω ότι μιλάμε μέχρι τώρα για κοινωνικέ και ιατρικέ ανταμοιβέ μόνον και όχι οικονομικού χαρακτήρα. Επίση, ε, θέλουμε να επιδιώξουμε πρότυπα ποιότητα για την επαγρύπνηση του συστήματο αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώ και την αποτελεσματική προστασία των δοτών. Η οδηγία δεν ορίζει ε, τι προδιαγραφέ για του δότε και του λήπτε, μόνο για τα όργανα τα ίδια και θα πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα στην οδηγία. Θα πρέπει να θίγει θέματα ποιότητα και ασφάλεια οδηγία, όπω το άρθρο 10 για την εχλασιμότητα και στο 11 για το σύστημα υποβολή εκθέσεων και τι σοβαρέ παρενέργειε. Όλα αυτά πρέπει να ενισχυθούν. Επίση, είναι σημαντικό να τονίσουμε για, ότι για όλες τις δωρεές η έννοια της ποιότητας και της ασφάλειας διαφέρει από ότι αυτή που εφαρμόζεται στα ίδια τα όργανα και τη μεταφορά τους. Εδώ έχουμε να κάνουμε περισσότερο με τη διαχείριση του κινδύνου σε επίπεδο μεμονωμένων ασθενών και λιγότερο σε σχέση με τον συνολικό κίνδυνο, όπως η πιθανότητα να μεταδοθεί κάποια ασθένεια. Η πατήτη δαγάμα ή κάποια ασθένεια ιολογικής προέλευσης. Έτσι λοιπόν η έκθεση του κυρίου Μικολάσιτ, όπω έχει προκύψει και από την έκθεση του κυρίου Πέρα Περαγιοροντίκη, δίνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν πολλέ κοινέ ιδέε, αλλά και κάποιε διαφορές μεταξύ των δύο σχεδίων έκθεση, όπω τις είδαμε σήμερα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε κυρίω την ερμηνεία τη αρχή τη μη αμοιβόμενη δωρεά και το ρόλο που θέλουμε να αναθέσουμε στου ζώντες δότες. Θέλουμε να προωθήσουμε την διδικασία αυτή ή όχι. Ίσως αυτό είναι μια τελευταία επιλογή. Και θα πρέπει να προβλέψουμε ένα σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη οργάνων. Βασικός παράγοντας που έχει πλήξει τα προγράμματα μεταφοράς. Εδώ να πω ότι πάνω απ' όλα δεν πρέπει να βλέπουμε τη μεταφορά ως ε, μια λύση αυτή καθ' αυτή. Θα πρέπει να είμαστε πολύ συνετοί αν θέλουμε να επιβάλλουμε την μεταφορά οργάνων, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ε, πλήγματα στην ισορροπία τη λειτουργία των συστημάτων δημόσια υγεία στο κατά μέλλον. Ευχαριστώ. Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. θα μιλήσω για την έκθεση Μικολάσιτς, γιατί μετά την επόμενη έκθεση χωριστά νομίζω θα τη συζητήσουμε. Η έκθεση του συναδέλφου Μικολάσιτς είναι πολύ σημαντική έκθεση. Μας ενδιαφέρει, γιατί ενδιαφέρει ως υπαρξιακό θέμα τους ανθρώπους. Θέλουμε να έχουμε ένα λογικό σύστημα που θα βοηθεί, θα βοηθάει τους ανθρώπους, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει εγγύηση για τις βασικές αρχές και αξίες. Πρώτο σημείο. Ε, θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι. Το 2008 είχαμε την έκθεση μου, είχαμε ε, ε, συζητήσει με την κυρία Μπρέπελς και καταλήξαμε σε κάποια σχετική συνένεση για το τι θέλουμε να κάνουμε με την οδηγία αυτή και είπαμε ότι θέλουμε μια οδηγία αλλά δεν θέλουμε υπερβολική γραφειοκρατία. Είχε φροντίσει ο εισηγητή λοιπόν πάρα πολύ επί του θέματος και ο πρόεδρος Γιώ Λάινεν ανέφερε και ένα άρθρο σχετικά με τη σημασία των αρχών ο κύριος ε, Μικολάσιτς στο άρθρο 18 καλά το χειρίζεται. Πρέπει να είναι ένας φορέας που θα έχει εξουσιοδοτηθεί από το κράτος μέλος. Μπορεί να είναι κάποια αρχή, μπορεί να είναι κάποιος οργανισμός, να είναι κάποιος φορέας, που θα πρέπει όμως να έχει την εξουσιοδότηση από το κράτος και θα πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγει ελέγχους. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι αυτή η αρμόδια αρχή. Νομίζω και από τα κράτη-μέλη είναι θετικά τα σχόλια που έχουμε πάρει επί του θέματος. Να συνεχίσουμε λοιπόν πάνω στη γραμμή που προτείνει ο κύριος Μικολάσης. Δεύτερο σημείο για την ιχνηλασιμότητα. Είναι κάτι που για τις λεπτομέρειες μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αν το όργανο πληγεί από κάποιο ιό, από κάποια μεταδοτική νόσο, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα ιχνηλασιμότητας. Μπορεί να είναι ένας ε, μεταθανάτιος ε, δότης και να διαπιστώσουμε εκ των υστέρων ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Μπορεί να, αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με έναν ασθενή ο οποίος δέχθηκε τη δωρεά, ήταν δότης του νεφρού, ήταν συγγνώμη λήπτης ε, του νεφρού, ε, ενώ πρέπει να αναζητήσουμε και τον λήπτη της καρδιάς από τον ίδιο μεταθανάτιο δότη, παραδείγματος χάρη, να ανακαλύψουμε κάποια μεταδοτική ασθένεια. Επ' αυτού λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε. Στα άρθρα 13 ε, και 16 έχουμε πολύ καλές προτάσεις από την Επιτροπή και προτείνει κάποιες βελτιώσεις ο κύριος Μικολάσης και σε αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουμε ώστε να έχουμε μια κοινή βάση Δεν ξέρω αν είμαστε πιο κοντά στην άποψη της Επιτροπής ή στην άποψη του κ. Μικολάσιτς. Θα δούμε και τι θέλουν και οι άλλες πολιτικές ομάδες. Πάντως, ενάντια του Συμβουλίου θα πρέπει να ενισχύσουμε το κείμενο, να μην το αποδυναμώσουμε. Η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου συνέταξε μία γνωμοδότηση για το άρθρο 13 και τμήματα του άρθρου 15, όπου λέει ότι δεν είναι συμβατά με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας. Παραβιάζουν την αρχή της επικουρικότητας και δεν συμφωνεί με την νομική τους βάση. Νομίζω ότι ε, έχει άδικο η νομική υπηρεσία. Δεν είμαι νομικός εγώ ίδιος, αλλά έχει νομική υπηρεσία και η Επιτροπή που εξήτασε αυτή την ε, νομοθετική πράξη πριν εκδοθεί. Το 2002-2003 είχαμε κάνει μια συζήτηση για την ποιότητα και την ασφάλεια ιστών και κιτάρων και είχε ε, τότε το Κοινοβούλιο την άποψη που έχει τώρα η Επιτροπή. Η Επιτροπή το έβλεπε τότε διαφορετικά, αλλά η δική μα νομική πάντοτε ήταν υπέρ αυτή τη κατεύθυνση. Δεν είμαι νομικό εγώ ίδιο, επαναλαμβάνω, αλλά ξέρω ότι και για αυτό το θέμα και για πολλά άλλα θέματα, αν ρωτήσει τρει νομικού, θα έχουν τρει διαφορετικέ απόψει. Γι' αυτό ε, είναι σαφέ ότι πρόκειται για ένα πολιτικό πρόβλημα εδώ. Τα κράτη-μέλη θέλουν ε, να δώσουν λίγε αρμοδιότητε, το δυνατόν λιγότερε αρμοδιότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σαφώ υπάρχουν ε, κάποια κράτη-μέλη τα οποία θέλουν να αφήσουν ανοιχτέ κάποιες, να αφήσουν ανοιχτά κάποια παραθυράκια. Μπορεί να μιλούν υπέρ της δυνατότητας δωρεάν οργάνων, δωρεάς οργάνων, αλλά αφήνουν ένα παραθυράκι για να μην είναι δυνατόν για διάφορους νομικούς λόγους να γίνει. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχει ενιαία θέση εδώ το Κοινοβούλιο, Μπορούμε να μιλάμε για θέματα λεπτομέρεια, αλλά δεν θα πρέπει να υπαναχωρήσουμε σε σχέση με την πρόταση τη Επιτροπή. Η πρόταση τη Επιτροπή είναι το ελάχιστο το οποίο θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε σε αυτά τα θέματα. Και δεν είναι μόνο θέμα ηθικής ή μόνο θέμα αρχών. Έχει σχέση με την ποιότητα και την ασφάλεια. Αλλά εδώ μιλάμε και για την τεχνική, τεχνική αναγνώρισης των ιών, ε, τεχνική σε σχέση με τις ε, ασθένειες. Και αν ένας δωρητής ε, πάρει 30.000 ευρώ ή 30.000 δολάρια για τη δωρεά, δεν έχουμε καμία εγγύηση ότι θα λέει την αλήθεια στον ε, γιατρό του ότι ε, προσέχει και δεν έχει σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα ή ότι δεν έχει κάποια άλλη ασθένεια. Κάποιους ιούς δεν μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε άμεσα και γι' αυτό η αρχή της ανοδιοτελούς δωρεάς είναι απόλυτη προϋπόθεση για να διασφαλίσουμε την ποιότητα και την ασφάλεια και για να εμποδίσουμε την μετάδοση ιών. Αυτή είναι η θέση του Κοινοβουλίου, αυτή είναι και η θέση της Επιτροπής και θα πρέπει κάπως περισσότερο να το διευκρινίσει η Επιτροπή. Στην πρόταση της Επιτροπής ίσως σε κάποια σημεία δεν εκφράζεται τόσο ξεκάθαρα και νομίζω ότι θα πρέπει να το εκφράσουμε ξεκάθαρα έναντι του Συμβουλίου. από την εμπειρία σε αυτό το θέμα και οι περισσότεροι συνάδελφοι θα το γνωρίσουν αυτό. Όταν κάποιος λέει ότι καταρχήν συμφωνούμε, αλλά για νομικούς λόγους διαφωνούμε, κάτι, κάποιος πολιτικός λόγος υπάρχει από πίσω και γι' αυτό είναι σημαντικό να ακολουθήσει μια αποφασιστική στάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ. Η πρόταση της Επιτροπής είναι το ελάχιστο πάνω στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε και να το βελτιώσουμε δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να περιοριστούμε σε κάτι χαμηλότερο από την πρόταση της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Λίζε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πριν από τέσσερις εβδομάδες... Είχα την ευκαιρία όταν ένας συνεργάτης μου ε, έγινε λήπτης οργάνου, ε, είδα πώς βελτιώθηκε η ποιότητα ζωής αυτής της συνεργατηδός μου. Έχω λοιπόν και μια προσωπική πρόσφατη εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, πολύ σοβαρό το θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να μας απασχολήσει ε, και σε λεπτομέρεια, αλλά να το προωθήσουμε και όσο το δυνατόν ταχύτερο. Ο εισηγητή νομίζω έχει προετοιμάσει μια πολύ καλή έκθεση. Ιδιαίτερα τονίζουμε το θέμα της ποιότητας και της ασφάλειας των οργάνων, που είναι πολύ σημαντικό και τονίζεται και στην τροπολογία 15 ε, και ε, σαφώς θα πρέπει ε, να μιλάμε για ιδιωτελεί δωρεά χωρίς αμοιβή. Δεν μπορεί να επαναχωρήσουμε στο σημείο αυτό. Ε, να μην υπάρχει δυνατότητα παρέκκλησης από αυτή τη βασική αρχή. Δεν είναι τόσο απλή βέβαια η κατάσταση και στην Ευρώπη έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα όσον αφορά τι δωρεέ οργάνων. Στην Ισπανία, παραδείγματο χάρη, υπάρχουν πολύ περισσότεροι δωρητέ από ό,τι σε άλλα κράτη-μέλη. Αλλά δεν θα πρέπει ε, να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα είναι λιγότερο προχωρημένο. Θα πρέπει ε, να ακολουθήσουμε ένα σύστημα που θα εγγυάται την υγεία και ε, την ασφάλεια. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία με την έκθεση αυτή. Και υποστηρίζω τον Πέτερ Λίζε που έλεγε το λόγο πριν από μένα, να μην επαναλάβω κι εγώ τα ίδια. Ας εγκρίνουμε λοιπόν την έκθεση αυτή το συντομότερο δυνατόν, γιατί όπως σας είπα έχω μια πρόσφατη εμπειρία και είδα πόσο ωραίο είναι να υποφελείται κανείς από μια δωρεά. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ρώση. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό. Το θέμα της ανωνυμίας, το οποίο έθιξαν αρκετοί συνάδελφοι, δεν είναι κατά την άποψή μου το πιο σημαντικό πρόβλημα. Σαφώς και είναι σημαντικό, αλλά όποιος είναι διατεθειμένος να ε, λάβει όργανα, ε, ή να δωρήσει όργανα έχουν ως βασικό πυλώνα την ανωνυμία τους. Αυτό θα πρέπει να είναι η κορονίδα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μία βεβαιότητα ποιότητας της έκθεσης Και νομίζω ότι προσπαθούμε να θέσουμε πολύ συγκεκριμένα όρια για τα χαρακτηριστικά του δωρητή, και επομένως των οργάνων τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται και μεταμοσχεύονται και χρησιμοποιούνται. Έχω δύο αμφιβολίες πολύ μικρές. Τροπολογία 31. Μιλάμε για δωρεές εν ζωή, οι οποίες ε, περιορίζονται ε, σε στενούς συγγενείς και συζύγους για να μην υπάρχει εκμετάλλευση. Ελπίζω να πρόκειται για λάθος στην Ιταλική μετάφραση, αλλά συνήθως όταν μιλάμε για συζυγούς μιλάμε για ε, ζευγάρια τα οποία είναι ε, παντρεμένα, αλλά εγώ νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε και για ζευγάρια τα οποία ε, συζούν, συμβιώνουν, διότι και πάλι μπορούν να χαρακτηριστούν ζευγάρι και είναι κρίμα όταν ε, χρησιμοποιούμε τον όρο σύζυγη να μην μπορούμε να συμπεριλάβουμε και αυτά τα ζευγάρια και να μην μπορούν να δωρήσει ο ένας ε, τα όργανα του στον άλλον. Τώρα, αυτό όλο με το περιορίζονται κλπ. κλπ ε, δεν συνάδει με αυτό που έχουμε στο σημείο 20. Στο σημείο 20, στο σχέδιο έκθεση, στο άρθρο 18, καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν το θέμα της δωρεάς ε, εν ζωή ε, ως συμπληρωματικό της δωρεάς ε, μεταν θάνατον. Και λέμε ότι θα πρέπει να περιορίζεται σε αυτή την περίπτωση μεταξύ συγγενών ή άτομα τα οποία συμβιώνουν ή είναι παντρεμένα μεταξύ τους και ταυτόχρονα λέμε ότι καλούμε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν την προώθηση της δωρεάς ε, εν ζωή. Ε, αυτά τα δύο σημεία δεν συνάδουν μεταξύ των. Μία άλλη παρατήρηση στο σημείο 32 όπου μιλάμε για την αποζημίωση. Εγώ συμφωνώ απολύτως ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό να πληρώνει κάποιο για ένα όργανο ή να μην κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να απαγορεύεται η εμπορία οργάνων. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι κίνδυνοι ελοχεύουν σε τέτοιες συναλλαγές αλλά εδώ μιλάμε για ε, πιθανή αποζημίωση ε, δωρεάς εν ζωή, η οποία θα περιορίζεται μόνο στις δαπάνες, για παράδειγμα ταξίδι, φύλαξη κλπ. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και ένα σημείο για την εγγύηση της ε, διατήρησης της θέσης εργασίας του, γιατί σε ορισμένες χώρες, στην Ιταλία μεν προβλέπεται αυτό, αλλά σε άλλες χώρες δεν ε, ε, γνωρίζω, ε, μιλάμε για αποζημίωση των δαπανών του λοιπόν, των εξόδων του, αλλά ε, να υπάρχει και μια διασφίληση ότι όταν κάποιος κάνει δωρεά οργάνων ε, εν τη απουσία του δεν θα χάσει τη θέση εργασίας του, είτε δουλεύει στο δημόσιο, είτε δουλεύει σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Ένα τελευταίο σημείο και ολοκληρώνω, το σημείο 33, και εδώ κατά την άποψή μου υπάρχει ένα λάθος, Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ε, έχουν υποστεί ζημίες Μιλάμε για παράδειγμα για λάθος. Ε, όταν έχουμε μεταμόσχευση για παράδειγμα οφθαλμού και τελικά γίνεται μεταμόσχευση νεφρού. Μιλάμε για κάτι πολύ περιορισμένο το οποίο καλύπτει μόνο τα έξοδα κάποιου για τη δωρεά. Εδώ πάμε κατά των ε, κείμενων κανόνων γιατί αν κάποιος λόγω λάθους υγείας έχει κάποια ζημία, ακόμα και αν ε, δεν ε, κάνει δωρεά οργάνου και πάλι θα πρέπει να γνωρίζετε μια αναπηρία γιατί πλέον έχει μια αναπηρία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, αν κάνουμε μία ε, τροποποίηση αυτής της μορφής, ουσιαστικά απαγορεύουμε σε αυτόν που κάνει δωρεά να λάβει την δέουσα αποζημίωση. Ή υπάρχει λοιπόν λάθος στη μετάφραση εδώ, ή θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή να το διορθώσει λιγάκι τέλος πάντων, γιατί αυτό ο οποίο κάνει τη δωρεά ε, ε, έχει κάποια περισσότερα να λάβει. Σαφώς το νοσοκομείο δεν έτυχε τη σωστή μεταχείριση. Χρειάζεται λοιπόν και την ανάλογη αποζημίωση. Και τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Διευθυντής κ. Ρης, εάν θέλει να απαντήσει στους συναδέλφους. Η κυρία Μπρονκό μάλλον. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή για τη δουλειά του. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Μικολάσιτ. Πραγματικά το θέμα αυτό φάνηκε ότι τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Έδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασμό και στις συζητήσεις και στη δουλειά μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν κύριε Μικολάσιτ. Και αναμένουμε να περάσουμε στα επόμενα βήματα της όλης διαδικασίας. Να θυμίσω ότι η Επιτροπή υπέβαλε αυτή την πρόταση μετά από μακρά διαδικασία διαβουλεύσεων και περίοδο μελέτης. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η Επιτροπή είναι να διαρθρώσει το κείμενο με μεγάλη προσοχή, ώστε να μην επηρεάσει υπάρχοντα συστήματα τα οποία ήδη λειτουργούν καλά. Να θυμίσω ότι η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 168. Επομένως, έχει κάποιους περιορισμούς που επιβάλλει στα ζητήματα που θα θέλαμε να καλύπτει. Δεν το επιτρέπει όμως κάτι τέτοιο νομική βάση. Αυτό είναι ένας τρόπος να εξηγήσουμε γιατί έχουμε οδηγία από τη μια και πρόγραμμα δράσης από την άλλη, που είναι το επόμενο σημείο στην ημερήσια διαταξή σας ούτως ή άλλως. Έτσι σημειώνουμε με μεγάλη ικανοποίηση ότι ο εισηγητής συμφωνεί με τις βασικές αρχές που περιλαμβάνει η πρότασή μας και ότι πολλές τροπολογίες απλώς σχετίζονται με κάποιες λεπτομέρειες στη διατύπωση. Για πολλές από τις προτινόμενες τροπολογίες διαβλέπουμε σύγκληση απόψεων μεταξύ Επιτροπής και Ευρωκοινοβουλίου. Όμως να τονίσω ότι για κάποια σημεία Ίσως κάποια από τα μέλη εδώ να έχουν ήδη αναφέρει τις ανησυχίες του σχετικά. Εκεί να τονίσω ότι μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για οδηγία. Η οδηγία, σε αντίθεση με έναν κανονισμό, αφήνει περιθώρια ευελιξία στα κάτι μέλη όταν μεταφέρεται και υλοποιείται. Εκεί να επιλέγουν πώς θα την μεταφέρουν και θα την υλοποιήσουν στην εθνική τους νομοθεσία. Κάποιες λοιπόν μικρές προσαρμογές μπορούν να γίνουν σε εκείνο το στάδιο ώστε να ληφθεί υπόψη η εθνική νομοθετική πραγματικότητα και το σχετικό πλαίσιο. Το σημείο το οποίο εγώ έχω εντοπίσει και ε, φαίνεται να ενδιαφέρει περισσότερο τους βουλευτές, αλλά να προκαλεί και τα περισσότερα σχόλια και ανησυχίες, είναι η οικειοθελής δωρεά. Αυτό που μπορέσαμε να αποδείξουμε μέσα από τη διαδικασία μελέτης και διαβουλεύσεων είναι ότι ο θελής και αμοιβόμενη δωρεά είναι ένα από τα κριτήρια το οποίο θα εγγυηθεί ασφάλεια και ποιότητα. Συμφωνώ ότι όπως έχει διατυπωθεί το κείμενο ίσως δεν τεκμηριώνει ούτε θεσπίζει ούτε απηχεί με κάποιον ρητό τρόπο την διασύνδεση αυτή. Όμως στην πραγματικότητα γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτή η διασύνδεση. Αυτό είναι και ο βασικός λόγος που στο άρθρο 168 και στην πρόταση που απορρέει από αυτό έχει αναφέρει την οικειοθελή αμοιβόμενη δωρεά η Επιτροπή. Τώρα τα παρεπόμενα πλεονεκτήματα της πρότασης αυτής είναι ότι γλιτώνουμε τον δότη από την ε, μη αναγκαία πίεση, την ανεπιθύμητη πίεση να λάβει αμοιβή για τη δωρεά. Επίσης καταπολεμούμε τη διακίνηση οργάνων, διότι δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο, δεν υπάρχει και λόγος να διακινούνται ανθρώπινα όργανα. Αυτή είναι η στόχη μας και έτσι γι' αυτό επιδιώκουμε την οικειοθελή αμοιβόμενη δωρεά. Τα σχόλια σε σχέση με την ιχνηλασιμότητα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ανησυχίες για τον τρόπο κατά τον οποίο θα επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία. Η Επιτροπή όμως πιστεύει ότι η πρόταση πραγματικά έχει ενσωματώσει την αρχή της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ προστασίας της ταυτότητας των δοτών και της ιχνηλασιμότητας σε περίπτωση ανάγκης. Άκουσα πολλοί να αναφέρουν περιπτώσεις όπου ο δότης εντοπίζεται βάσει της ηλικία του. Καλό θα ήταν λοιπόν να μπορούμε να εντοπίσουμε εφόσον το θέλουμε και τους λήπτες των οργάνων. Να αναφέρω και να σας θυμίσω ότι ένας ε, δωρητής οργάνων μπορεί να είναι και δότης ιστού. Αυτό θα επηρεάζει πολύ περισσότερους ασθενείς από ότι τους λήπτες ε, γλώσσα, νεφρών, ε, σηκωτιού και άλλων οργάνων. Αυτό για μας λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και το σκεφτήκαμε διαμακρών, επί πολύ καιρό μέχρι να καταλήξουμε σε μια σωστή και ισορροπή λύση. Ίσως να υπάρχουν καλύτερες διατυπώσεις από αυτές που πρότεινε ο ελεγκτής για την ασφάλεια των δεδομένων, αλλά αυτό θα το επεξεργαστούμε. Μπορούμε πάντως να το λάβουμε υπόψη για την επαναδιατύπωση που θα γίνει Επίσης η Eurotransplant. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όπως κάνουμε ως τώρα. Και όλοι αναγνωρίζουμε ότι το έργο που γίνεται ως τώρα είναι εξαιρετικό. Η πρόταση όμω διατυπώθηκε, όπως είπαμε, ιδιαίτερη προσοχή για το άρθρο 22, στοχεύει ακριβώς να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν εμπόδια στην εξακολούθηση της δράσης των συστημάτων όπως του γεροτρανσπλαντ. Απευθύνθηκε έκκληση για μια κάρτα Ευρωπαίου δόρητη. Νομίζω ότι ήδη στην εισαγωγή μου το συζήτησα αυτό και κάλυψα το ζήτημα της νομικής βάσης. Εδώ αυτό ξεπερνά τα όρια που μας επιτρέπει η νομική βάση, το άρθρο 168. Το γεγονός ότι δεν έχουμε μια για τη δωρεά οργάνων στα διάφορα κατημέλη μέλη είναι κάτι που όλοι το παραδέχονται. Άκουσα επίση έκκληση από κάποιον ότι θα πρέπει να διδαχθούμε από τι πρακτικέ που χρησιμοποιούνται στα διάφορα κράτη-μέλη. Δεν θέλω να προκαταλάβω το επόμενο σημείο στην ημερήσια διαταξή σα, όμω υπάρχει και το πρόγραμμα δράση που ακριβώ αυτό στοχεύει. Εάν μάλιστα μου δοθεί ευκαιρία στη συζήτηση για το επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, θα φροντίσω να παρέμβω. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ σα ευχαριστώ. Κύριε Σιγητά, Θέλετε κάτι να προσθέσετε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ όλους γιατί λάβατε μέρος σε αυτή τη συζήτηση και για τα σχόλιά σας στην έκθεση αυτή. Σημειώνω όλες σας τις ανησυχίες, όλα σας τα σχόλια. Ε, καλό θα ήταν να μην ε, παρατείνουμε τη συζήτηση για σήμερα. Θα φροντίσω να συνεργαστώ μαζί με όλους εσάς και σε διμερές επίπεδο για να φροντίσω να συμπεριλάβω όσο το δυνατόν περισσότερο τις παρατηρήσεις σας στο κείμενο, να γίνουν σχετικές προσαρμογές και να έχουμε και το χρόνο να εξεύρουμε μια καλύτερη διατύπωση ή να απηχηθεί το περιεχόμενο των δικών σας παρατηρήσεων, αλλά και να μείνουμε πιστοί στο πνεύμα της οδηγίας. Το κείμενο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να το υπερασπιστούμε, διότι είμαστε το κοινοβούλιο, είμαστε βουλευτές. Πρέπει να δείξουμε με κάθε τρόπο ότι συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση και να περάσουμε ένα μήνυμα ηχηρό ότι ο τομέα αυτός μας ενδιαφέρει. Η Ευρώπη χρειάζεται πιο πολλά όργανα, πιο πολλέ μεταμοσχεύσεις. Συμφωνούμε εδώ λοιπόν όλοι από ό,τι φαίνεται ότι αυτό είναι ο λόγος που κάνουμε αυτή τη δουλειά και καλώ κάνουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Πολύ σύντομα μόνο να σχολιάσω την παρατήρηση του κυρίου Ρώση. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια παρανόηση. να είστε βέβαιος ότι εδώ δεν είναι θέμα ουσίας αυτό που σας απασχολεί, αλλά μορφής. Επίσης, να μην ξεχνάμε και την αντεχόμενη ζημία του προσώπου που είναι ζών δότης, γιατί ο κύριος Λίζε που είναι γιατρός και η συνάδελφος που μίλησε προηγουμένως ξέρουν ότι ο δότης μπορεί να έχει ιατρικές επιπλοκές μετά τη δωρεά. Αυτό λοιπόν ήθελα να καλύπτεται εδώ. Αυτή ήταν η μεριμνά μου. Να έχει κανείς την ευγένεια να δορίζει το όργανό του και μετά να γνωρίζει επιπλοκές, να μπορεί να λάβει κάποια αποζημίωση. Και μετά θα συμφωνήσουμε για τη διατύπωση σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Φαντάζομαι ότι ούτως ή άλλως στην ουσία συμφωνούμε. Λογικό είναι να θέλουμε μια πιο ανθρώπινη, μια προσωποπαγή προσέγγιση. Ευχαριστούμε λοιπόν, ευχαριστούμε και την Επιτροπή, την οποία ότως ή άλλως συνείδησα κατά την αρχή των εργασιών μου και τους ευχαριστώ για τον υποδομητικό τρόπο συνεργασίας που είχαμε. Θα χαρώ να συνεργαστώ μαζί σας και στο μέλλον και πραγματικά χαίρομαι που το κείμενο σας απασχολεί, που υποβάλλετε συνεχώς παρατηρήσεις ώστε να καταλήξουμε σε ένα άριστο κείμενο το Μάρτιο στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής και μετά να δούμε την ε, συμφωνία της πρώτης ανάγνωσης τον Απρίλιο και στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Ευχαριστώ. Κύριε Μικολάση, σας ευχαριστώ για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, η ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 11 Φεβρουαρίου 2010, αλλά θα ακολουθήσουμε μια νέα διαδικασία σε αυτή την περίπτωση που θα μας επιτρέψει, θα επιτρέψει στους ε, βουλευτές και στους όσους μπορούν να υποβάλουν τροπολογίες να τις αποβάλουν online στο διαδίκτυο. Τώρα, για το πώς θα γίνεται ακριβώς αυτό από τεχνικής άποψης, θα χρειαστούν μάλλον λίγες ώρες ε, κατάρτισης για όσους θα προτιμήσουν αυτή τη μέθοδο. Τέλος πάντων, για τη νέα αυτή μέθοδο και για την Επιτροπή Περιβάλλοντος που δεν την έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ πριν, έχει γίνει αυτό σε άλλες επιτροπές, αλλά όχι αυτήν. Για αυτό το κείμενο λοιπόν ακριβώ θα την πρώτο χρησιμοποιήσουμε. Θα ανασκομποθούμε και θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη διαδικασία. 16 Μαρτίου λοιπόν στην Επιτροπή ψηφίζουμε και τον Απρίλιο στην Ολομέλεια. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, σημείο 20. Δίνω το λόγο στον κύριο Περέγιο για την έκθεσή του για το ζήτημα που ακριβώς συμπληρώνει αυτό που μόλις συζητήσαμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αν έπρεπε να δώσω έναν ε, πρακτικό και απλό ορισμό, με τον κίνδυνο να είμαι πολύ απλουστευτικός, ε, να πω ότι το κείμενο το οποίο θα σας παρουσιάσω, κατά την άποψή μου, είναι το συμπλήρωμα για την καλή εξέλιξη και εφαρμογή της οδηγίας τόσο για να καθοριστεί το πρόγραμμα αυτό, αλλά και γιατί ε, κάποια στιγμή θα πρέπει να το αξιολογήσουμε αυτό με στην ευρωχόμενη πενταετία. Όπως γνωρίζετε, ε, το κείμενο σας είναι λίγο πολύ γνωστό, γι' αυτό λοιπόν δεν θα το εξηγήσω παράγραφο προς παράγραφο, θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις, ε, κάποιες γενικές ε, παρατηρήσεις για αυτό που συζητάμε για να μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση δεδομένου ότι έχει περάσει και η ώρα. Προσπαθούμε να έχουμε συνεργασία μεταξύ κρατών μελών ε, ορίζοντας κάπως το συντονισμό δράσεων και καθορίζοντας κοινέ. Ε, ε, κατευθυντήριες γραμμές και για να αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων οργάνων προς μεταμέσχευση ε, αλλά και για το ε, γεγονός ότι, να το υπενθυμίσω, το ξέρω ότι επαναλαμβάνομαι συνεχώς, αλλά ε, δυστυχώς ε, είναι πάρα πολύ λίγα τα όργανα. Υπάρχουν σχεδόν 100.000 άτομα στην Ευρώπη που περιμένουν στη λίστα αναμονή για τη δωρεά ενός οργάνου και είναι σχεδόν δύο την ημέρα τα άτομα τα οποία όντως λαμβάνουν αυτό το όργανο και μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους. στα διάφορα εκτιμώντες ε, του κειμένου εξηγούνται αρκετά καλά ε, δύο βασικοί στόχοι που θεωρώ ότι υφέρπουν σε όλο το κείμενο και ε, θα ήθελα να τους επισημάνω αν δεν τους διαπιστώνετε γραπτός. Ο στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ε, απλή ε, και στο θέμα των μεταμοσχεύσεων. Να, και πώς θα γίνει αυτό, συντονίζοντας τα πράγματα, συνειδητοποιώντας ότι όλοι είμαστε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό θα πρέπει να γίνει όπως και σε πολλά άλλα θέματα και για τις μεταμοσχεύσεις. Ε, δεν θα σας δώσω τα εθνικά στοιχεία, αλλά θέλουμε να διαψεύσουμε αυτό τον μύθο, ο οποίος κατά την άποψή μου είναι λανθασμένο, των χωρών που προστατεύουν μόνο τους εαυτούς τους. Ε, θα σας μιλήσω λοιπόν για το λανθασμένο μύθο της Ισπανία. Δεν είναι αλήθεια ότι εμείς είμαστε πιο αλληλέγγυοι από την υπόλοιπη Ευρώπη, διότι βάσει των τελευταίων στοιχείων που διαθέτουμε, τουλάχιστον 13 χώρες όταν τους ε, ε, ρωτάνε αν ε, θέλουν να κάνουν δωρεά οργάνων, βρίσκονται πάνω από, την Ισπανία σε χώρες δωρητές. Δεν είναι αλήθεια λοιπόν ότι η Ισπανία είναι πιο αλληλέγγυα από τους υπολείπους. Τι γίνεται είναι ότι... Στην Ισπανία έχουμε 35 περίπου τις 100, ενώ στην Βουλγαρία έχουμε 1,1%. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δίνονται από τα στατιστικά δεδομένα και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και γιατί εμφανίζονται έτσι τα ποσοστά. Αφενός ε, γιατί η παιδεία στο θέμα των μεταμοσχεύσεων, τόσο σε αφορά στους επαγγελματίες όσο και στους πολίτες, ε, είναι πολύ άνηση. Σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ανύπαρκτη. Τα εθνικά συστήματα λειτουργούν με άνισο τρόπο και άνισες δομές και ακριβώς ε, δεν υπάρχει ένα μέσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που μας επιτρέπει να συντονιστούμε και να έχουμε πιο ευέλικτα και πιο αποτελεσματικά συστήματα για κοινό συντονισμό στο κείμενο ε, αναφερόμαστε στην εγγύηση και στην ασφάλεια των οργάνων, την ε, κατάλληλη κατάρτιση των επαγγελματιών. Είναι πολύ απαραίτητη η συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωση των επαγγελματιών στα νοσοκομεία. Γι' αυτό μιλάμε για νοσοκομιακό προσωπικό ή κέντρο υγείας που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Καθώς επίσης και να υπάρχουν και άτομα στα νοσοκομεία που ε, αντιμετωπίζουν με ευαισθησία τα θέματα που θέτουμε εδώ στο ε, κείμενο αυτό. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε να ε, επισημαίνουμε συνεχώς ε, το ρόλο των των δωρεών, όχι μόνο ως εγγύηση, αλλά και γιατί θεωρούμε ότι είναι η συλλογική εγγύηση που χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το εν λόγω ζήτημα. Ε, προσπαθούμε να επιμηκύνουμε τη ζωή κάποιου, ξεκινώντας από την αλτρουιστική δωρεάν, ε, δωρεά ενός οργάνου, Και όταν μιλάμε για το θέμα αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς. Εμείς ε, στο σχέδιο κειμένου λέμε ότι δεν αποκλείεται η αποζημίωση των δαπανών ε, κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης, αλλά πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι αυτή η έννοια, όπως θέλετε αποκαλέστε την αποζημίωση, καταβολή εξόδων ή οτιδήποτε, ε, δεν έχει καμία σχέση με τη δωρεά αυτή καθεαυτή, διότι αυτός που δωρίζει ένα όργανο δεν περιμένει τίποτα παραπάνω παρά ευγνωμοσύνη από αυτόν που του δώρισε το όργανό του, ε, ένας άνθρωπος ο οποίος ε, μπορεί να ήταν θύμα ενός ατυχήματος ή οποιασδήποτε άλλης ε, πάθησης. Να σας πω ότι το κείμενο, το λέω και ως πάντα μπορεί να βελτιωθεί και το κατανοώ ότι μπορεί να βελτιωθεί όχι μόνο για την ουσία του, γιατί ε, σαφώς ε, κάποιες ε, βελτιώσεις ε, θα προτείνω και εγώ ο ίδιος ως εισηγητής μέσω τροπολογιών, αλλά ε, και οι σκιώδες εισηγητές ε, με βοήθησαν με ένα διάλογο και ξέρουμε όλοι ότι μπορεί να χρειάζεται καλύτερη διατύπωση, καλύτερη μορφή σε κάποια σημεία. Οποιαδήποτε πρόταση γίνει για να βελτιώσουμε το κείμενο, για να έχουμε καλύτερο συντονισμό με την οδηγία και να έχουμε και οτιδήποτε συμπλήρωμα είναι ε, καλό για την εξέλιξη της οδηγίας, το είπα και από πριν, ε, πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Και εδώ συμφωνώ με όλους όσους το είπαν αυτό. Υπάρχει όμως η δυνατότητα αυτή και η δυνατότητα για βελτιώσεις είναι πάντα ευπρόσδεκτη, διότι πρόκειται για ένα σχέδιο κειμένου, το οποίο μπορεί με να μην είναι εκτενές, αλλά ουσιαστικά η πρόταση που κάνει είναι πολύ ευαίσθητη και θα πρέπει να το εξετάσουμε με την ανάλογη ευαισθησία. Ε, το να είναι κάτι δωρεάν, το να υπάρχει εμπιστοσύνη, να μην καταβάλει κάποιος τα έξοδα. Ε, όλα όσα προέκυψαν εδώ και είναι σημαντικά για όλους. Και νομίζω ότι και στο προηγούμενο ε, θέμα όσοι όσοι παρενέβησαν είχαν ένα κοινό στόχο και αυτό το στόχο προσπαθώ να προσπίσω και εγώ. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λίζα. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Πίτερ Λίζα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Περίγιο για την πολύ καλή, τον συνάδελφο Περέγιο για την πολύ καλή έκθεση. Όπως είπα και στην Υπουργό, έτσι και ο κύριος Περέγιο είναι Ισπανός, που είναι από χώρα πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο. Πρωταθλήτρια όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στη δωρεά οργάνων. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Ισπανοί είναι πιο πρόθυμοι να προβούν σε δωρεά οργάνωση σε σχέση με άλλους πολίτες, αλλά είναι καλύτερα οργανωμένο το σύστημα δωρεάς στη χώρα μου. Υπάρχουν όργανα τα οποία δεν ε, λαμβάνονται παρότι οι ε, δότες έχουν ταυτότητα ε, δότη. Και κατά τη γνώμη μου αυτό αποτελεί ένα τεράστιο σκάνδαλο και σε πολλές χώρες υπάρχει πρόβλημα ε, ε, στο σύστημα. Κανείς δεν είναι έτοιμος να οργανώσει το σύστημα σωστά. Και δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους γιατρούς. Ένας γιατρός σε ένα νοσοκομείο προσπαθεί να σώσει τη ζωή των ανθρώπων και δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν με έναν αποθανόντα δότη από τον οποίο θα μπορούν να λάβουν, να αφαιρέσουν πιθανά όργανα δωρεάς. Γι' αυτό χρειάζεται ένας συντονιστής δωρεάς. Γιατί πολύ συχνά ε, η δωρεά οργάνων εξαρτάται από αυτό το συντονισμό. δεν είναι ε, σημαντικό το αν έχουμε ένα σύστημα άρνησης ή ένα σύστημα έγκρισης ε, όσον αφορά ε, την συνένεση και την εξουσιοδότηση. Πιστεύω ότι το σύστημα οργάνωσης είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε. Η έκθεση αποτελεί μια καλή βάση και θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε παραπάνω και όπως ε, και στην έκθεση Άνταμο του 2008 ε, θα πρέπει να εξετάσουμε τη διατύπωση ούτως ώστε να είναι πιο ευανάγνωστη η έκθεση και το ένα κεφάλαιο να ακολουθεί το προηγούμενο. Υπάρχει ένα πολύ ευαίσθητο σημείο με πολλές αντιφάσεις ε, το θέμα των ενζοή δοτών. Οι ενζοή δότες θα είναι ένα κεφάλαιο συμπληρωματικό Πάντοτε είναι προβληματικό το θέμα των ενζοειδωτών και θα σας δώσω ένα παράδειγμα από τη Γερμανία. Πριν από λίγα χρόνια ήμουν σε μια κλινική και υπήρχε ένας πολίτης από το Ισραήλ που είχε πει ότι ήταν με ένα, με ένα συγγενή του που είπε ότι έρχεται από την Μολδαβία. Τελικά η αρμόδια αρχή αρνήθηκε τη δωρεά αυτή γιατί ήταν σαφές ότι πρόκειτο περί δωρεάς επαμοιβή, δεν ήταν πραγματική συγγενής με τους εν ζωή δότες, αν δεν υπάρχει πραγματικά στενή σχέση και αν απλώς δηλώνουν ότι πρόκειται για θελοντές δότες, πολύ συχνά ε, παραβιάζεται η αρχή της ανιδιοτελούς δωρεάς. και στο 17, στην παράγραφο 17 μιλάμε για διευρυμένα κριτήρια. Ε, παλιότερα λέγαμε ότι μετά τα 60, μετά τα 70 δεν μπορούμε να κάνουμε δωρεά. Τώρα πλέον από ιατρικής πλευράς δεν ισχύει αυτό. Μπορούμε να δώσουμε το, ένα όργανο από έναν, από έναν δότη 70 χρονών σε κάποιον άλλον 70 χρονών που περιμένει το συγκεκριμένο όργανο για μεταμόσχευση. σε πολλά κρατημέλη είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα των εν Μιλάμε για τον εγκεφαλικό θάνατο ως κριτήριο για την ε, δωρεά οργάνων. Ε, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε σε όλα τα επίπεδα για ε, τους εν και τους μεταθανάτιους δότες. Ο εισηγητής ε, μιλά επίσης ε, για την εμπορία οργάνων και για τον τουρισμό ε, σε τρίτες χώρες για απόκτηση οργάνων στην παράγραφο 24. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να προτείνονται και κάποιες κυρώσεις και ξέρω ότι στην Ισπανία ήδη συζητείται αυτό το θέμα. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην επιβαρύνουμε τους ασθενείς. Όταν ασθενείς, ε, παραδείγματος χάρη, ταξιδεύουν στην Ινδία για την απόκτηση ενός οργάνου θα πρέπει να συνεχίσουμε να τους θεωρούμε ασθενείς αλλά σαφώς να είναι, σαφέ, να είναι ξεκάθαρο ότι ε, είναι παραβίαση κάποιων ε, αρχών και επομένως είναι παράνομο. Ορισμένα ασφαλιστικά ταμεία προτείνουν στους ασθενείς τους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και να αγοράσουν ουσιαστικά ένα όργανο από κάποιο δότη εκεί, κάτι το οποίο δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχουν πολλές προτάσεις ε, που θα μπορούσαμε να κάναμε εν είδη τροπολογίας και το Μάιο ε, γίνεται μια συζήτηση στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ε, για το εμπόριο οργάνων και η Ευρώπη θα πρέπει να έχει μια σαφή θέση. Και εδώ νομίζω ότι και η Europol θα πρέπει να μας ε, υποστηρίξει γιατί ε, πρέπει να ασχολείται η Europol με αυτό το θέμα. Είναι καθήκον της Europol να διερευνά τέτοια θέματα. Έχουμε θέσει το ερώτημα στα κράτη-μέλη αν υπάρχει εμπόριο οργάνων η απάντηση των κρατών μελών ήταν όχι, επομένως η τελική διαπίστωση ήταν όχι, δεν γίνεται εμπόριο οργάνων. Όμως, σύμφωνα με δημοσιογραφικές ε, πληροφορίες, υπάρχει εμπόριο οργάνων και στα 27 κράτη-μέλη και μπορεί να μην γίνεται η μεταμόσχευση στα κράτη-μέλη, αλλά γίνεται η διαμεσολάβηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το εμπόριο οργάνων. Η Europol απέκλεισε αυτή την δυνατότητα και αυτό με λυπεί ιδιαίτερο. Θα έπρεπε η Europol να έχει περισσότερε πληροφορίε από το Συμβούλιο τη Ευρώπης ή από δημοσιογράφους. Η Europol είναι μια αστυνομική οργάνωση και θα έπρεπε να ασχολείται με αυτά τα οποία ε, ε, γίνονται κρυφά και όχι μόνο επιφανειακά να ρωτάνε ποιο έχει δηλώσει εμπόριο οργάνων, κανείς άρα δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν θα είναι κάτι στο, για το οποίο θα κάνουμε έκκληση στη Europol να ασχοληθεί πολύ πιο σοβαρά από ό,τι μέχρι τώρα. Ε, με μεγάλη μου χαρά περιμένω τη συνεργασία με τον εισηγητή και τους υπόλοιπους όδης εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πίτερ Λίζε. Κυρία Παρβάνοβα. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη ακούσα πάλι προσωπώ την ε, σκιώδη συγκεκριά μα, την κυρία Ρίζ, και να πω ότι προτείνει οι δύο εκθέσεις να θεωρηθούν ως ένα σύνολο. Θα μπορούσαν κάποιες από τις ιδέες τους να εξεταστούν από κοινού. Μην επαναλάβω λοιπόν τα ίδια που είπε προηγουμένως, απλώς ένα τελικό σχόλιο για όσους δεν είναι επαγγελματίες ιατροί. Όταν μιλάμε για ζώντες δότες, σε αυτή την περίπτωση δεν σημαίνει ότι καταλήγουμε μετά την παρέμβαση, την επέμβαση μάλλον σε δύο ε, ανθρώπους ε, με το ίδιο προσδόκιμο ζωής. Ο λήπτης ίσως να έχει τελικά μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής από ό,τι θα είχε προηγουμένως, αλλά όχι πάντοτε. Κάποιες φορές ο λήπτης αποβάλλει το όργανο. Και στο τέλος της ζωής τους λαμβάνουν ε, ειδικά φάρμακα για το ανοσοποιητικό σύστημα που επηρεάζουν ιδιαίτερα την υγεία τους. Το όργανο λοιπόν από ένα ανθρώπινο σώμα που μεταμοσχεύεται σε ένα άλλο σώμα σαφώς επηρεάζει τη ζωή του δότη, τον οργανισμό. Αυτό είναι ιατρικό το σχόλιο και πρέπει να το έχουμε πάντοτε κατά νου. γιατί μπορεί να υπάρχει ευκαιρία εδώ και δεν μιλάω για το νομικό σύστημα, αλλά το οργανωμένο έγκλημα κατά τη διακίνηση οργάνων. Ευρωπαίοι ασθενεί θα πάνε για τη μεταμόσχευσή του στο Πακιστάν. Και ένα πολύ συνηθισμένο προορισμό αυτό. Η πακιστανική κυβέρνηση επέβαλε πολύ αυστηρού κανόνε πρόσφατα για να εμποδίσει αυτή τη διακίνηση. Και υπάρχει και ένας παράνομος διάβλος οργανωμένου εγκλήματος για την παροχή σε λήπτες, παροχή οργάνων σε λήπτες. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε τις δράσεις αυτές με μεγάλη προσοχή, να είμαστε πολύ αυστηροί και να μην ενθαρρύνουμε τέτοιου είδους πρακτικές που είναι τελείως εγκληματικές. Ε, Ευχαριστούμε κυρία Μπρόνκο από την Επιτροπή. Thank you, Madam. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Εγώ θεωρώ ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ θετική για το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως σας είπα και προηγουμένως, πρόκειται για ε, συμπληρωματικό τμήμα της προτινόμενης οδηγίας. Το πρόγραμμα δράσης, το οποίο θετήθηκε στο τέλος του 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Και το ίδιο το πρόγραμμα δράσης εστίαζε σε 10 πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες, όπου οι συζητήσεις με τα κράτη-μέλη θεωρήθηκε ότι μπορούν να έχουν ένα επιπρόσθετο όφελος. Επομένως εστιάζουμε σε πολύ συγκεκριμένε δράσεις, ανταλλαγής πληροφοριών, οργανωτικές πτυχές, όπου τα κράτη-μέλη μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες και να βελτιώσουν την ε, κατάστασή τους και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν που κάναμε είναι να πάρουμε αυτές τις 10 προτεραιότητες ε, ε, τις οποίες τις έχουμε υποδιαιρέσει σε υποπροτεραιότητες για να μπορούμε να τις διαχειριστούμε πιο εύκολα και αυτή τη στιγμή συζητάμε και ε, ακούμε τι έχουμε να πούμε για τους δείκτες, διότι δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε την επίδραση ενός προγράμματος ε, δράσης αν δεν έχουμε κοινού δείκτες. Αυτές λοιπόν είναι οι κοινέ δράσεις που ξεκινήσαμε το 2009. Συζητήθηκαν επιπλέον δύο πτυχές το 2009 και θεωρούνται πάρα πολύ σημαντικές και ε, πτυχές ε, οι οποίες θα φέρουν ωφέλη πολύ γρήγορα. Πρώτον, οι οργανωτικές πτυχές και να προσπαθήσουμε να μεταλαμπαδεύσουμε τις παραδόσεις ή την ύπαρξη ε, μεταμοσχεύσεων σε κάποιες χώρες. Άκουσα σήμερα αρκετές φορές το θόμα της οργάνωσης, ε, το έθιξαν αρκετοί. Ε, το γεγονός ότι υπάρχουν όργανα αλλά χάνεται ευκαιρία να ε, μεταμοσχευθούν κάπου. Επομένως, το 2009 ε, ήταν προτεραιότητα το, το θέμα της οργάνωσης και θα συνεχίσει και για το 2010. Ένα άλλο στοιχείο ήταν ε, η κατάρτιση των εκπαιδευτών. Εκπαιδεύουμε ανθρώπους που αργότερα θα δείξουν στα, ε, στα νοσοκομεία συγγνώμη, πώς θα εφαρμόζεται καλύτερα το σύστημα. Έχουμε τακτικές συνεδριάσεις με τα κρυάτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα σταματήσει αυτή η διαδικασία, να διατηρήσουμε αυτή την ορμή που έχουμε λοιπόν Λοιπόν, και κάνουμε τακτικές συνεδριάσεις. Μια άλλη προτεραιότητα για το 2010 είναι να ανταλλάσσουμε πληροφορίες για προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας. Τα κράτη-μέλη που έχουν τέτοια προγράμματα μας έδωσαν την τεκμηρίωση και τις πληροφορίες που έχουν και το μοιραζόμαστε με τα άλλα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα νοσοκομεία στα οποία μπορούμε να εντοπίσουμε δωρητές και στα νοσοκομεία στα οποία γίνονται μεταμοσχεύσεις. Θα ήθελα να απαντήσω και σε ένα σχόλιο το θέμα της Europol. Εξ όσων γνωρίζω, η Europol, ή αν θέλετε η αστυνομία, έχει την αξής ε, διαδικασία εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει επίσημη ένσταση από κράτο μέλο πριν ξεκινήσει μια έρευνα. Πρόκειται λοιπόν για μια αστυνομία δεύτερη τάξεω, αν θέλετε, και εξ όσων γνωρίζουμε ποτέ δεν έχει γίνει τέτοια επίσημη ε, αίτηση για έρευνα. Όσον αφορά τώρα τη διακίνηση, να σας ε, διαβεβαιώσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες ποινές και υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο προσφάτως υιοθέτησε μία αναθεώρηση της απόφασης πλαίσιο για την καταπολέμηση της ε, διακίνησης ε, ανθρώπων, της εμπορίας ανθρώπων και το θέμα της εμπορίας οργάνων συμπεριλαμβάνεται ρητός ε, στο κείμενο. Επομένως υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον για την διακίνηση οργάνων. Το τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να θίξω για το πρόγραμμα δράσης είναι ότι θα γίνει μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση το 2012 του προγράμματος δράσης, γεγονό που θα μας επιτρέψει κατά τη δεύτερη περίοδο του προγράμματος δράσης να διορθώσουμε τυχόν προσανατολισμούς που θεωρούμε ότι ήταν εσφαλμένοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Σιγητά, έχετε κάτι να προσθέσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους κοιόδης ηγητές και τον κύριο Λύση και την κυρία Παρβανόβα. Το τόνος και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων τους ήταν σαφέστατος και να τους διαβεβαιώσω ότι για να μπορέσει να συνεχίσει το θέμα θα πρέπει να υπάρχει διάλογος που θα μας οδηγήσει να καταλήξουμε σε συμφωνία. Το θέμα που έθεσε ο κύριος ε, Λίζε το έθεσα και εγώ όταν συζητούσαμε την οδηγία θα πρέπει να γίνει σωστή διασύνδεση μεταξύ των δύο εγγράφων, την οδηγία και το πρόγραμμα δράσης και έτσι απαντώ και στην κυρία Παρβανόβα. Πρέπει να γίνει μια διαδικασία συντονισμού αυτών των δύο διαδικασιών, διότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού. Σε κάποια από τα σημεία Μιλάμε για διευρυμένα κριτήρια που μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε λίγο καλύτερα την προέλευση των οργάνων για να διασφαλίζουμε ότι δεν είναι από άτομα άνω των 70 ετών και είναι λογικό να θεωρούμε ότι το βέλτιστο είναι να έχει ο 30 με 35, ε, να είναι 30 με 35 ετών και αν κάποιος είναι πολύ μεγαλύτερη ηλικία θα είναι πολύ δύσκολη η μεταμόσχευση. Καλό είναι να γίνεται μεταξύ ατόμων αντίστοιχη ηλικία για να μπορέσουμε να έχουμε πολύ καλύτερε δυνατότητε μεταμόσχευση. Να πω επίση ότι όλα όσα κάνουμε προχωρούν και το είπε πολύ σωστά ο κύριο Λίσε, ε, γίνονται για να μην χανεί ούτε ένα όργανο διότι δεν υπάρχει συντονισμός, γιατί δεν υπάρχουν μέσα και γιατί η οικογένεια μπορεί δεν ξέρει να, να μην ξέρει να αναλύσει τη διάθεση του δωρητή και από κάποιες μικρολεπτομέρειες ορισμένες φορές χάνεται ένα όργανο και χάνεται μια ακόμα ζωή στην Ευρώπη. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε μέχρι να επιτύχουμε όλοι, διότι αυτή η επιτυχία θα είναι και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Euh, σα ευχαριστώ κύριε Σιγητά, για την ε, ποιότητα τη εκθεσή σα και για τι παρεμβάσει σα. Όπω και την προηγούμενη έκθεση, οι τροπολογίε μπορούν να κατατεθούν ω τι 11 Φεβρουαρίου το μεσημέρι με την ίδια διαδικασία. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μα θα γίνει στι 16 Μαρτίου 2010 και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Περνάμε τώρα στο προφορικό ερώτημα, προφορική ερώτηση μάλλον, τη κυρία Ριβαζή Κυρία Ριβαζή, έχετε το λόγο. Τι θα απαντήσει η Επιτροπή πριν την ερώτηση. Bon, donc... Euh, Πολύ ωραία. Να δώσω τότε το λόγο πρώτα στην Επιτροπή για να απαντήσει στην ε, γραπτή ερώτηση της κυρίας Ριβαζή και μετά θα μπορέσετε να συμπληρώσετε με άλλες ερωτήσεις αν το θέλετε κυρία Ριβαζή. Παρακαλώ. Ο αρμόδιος της Επιτροπής, ο κύριος Ρης. Κύριε Δευθυντά, έχετε τον λόγο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Η ερώτηση της κυρίας Ριβαζή γύρει διάφορα ζητήματα για την πανδημία H1N1. Τα μέτρα κατά του ιού όπω ελήφθησαν από τα κάτι μέλη για να αντιμετωπίσουν τις ε, δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας, με οδηγούν στο να σας παρουσιάσω μια συνολική εικόνα για το πώς διαχειριστήκαμε το θέμα αυτό. Δεν ήταν απλό. Λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος. Η πανδημία όμως αυτή εξακολουθεί να διαδίδεται και να εξαπλώνεται εδώ και νέα μήνες βάσει και η αντίδραση των, θε... των θεσμικών οργάνων, του κοινού, των δημόσιων φορέων ήταν πολύ καλή. Πολλοί από αυτού 24 ώρε το 24ωρο, 7 ημέρε την εβδομάδα προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Πολλέ λοιπόν ευχαριστίε σε όλου αυτού του ανθρώπου που φρόντισαν να καταπολεμηθεί η πανδημία. Από, την, από το πρώτο κρούσμα στο Μεξικό, από την αρχή της πανδημίας, η Επιτροπή αύξησε το επίπεδο επαγρύπνησης και ειδοποίησε τα κράτη-μέλη. Χάρη στην Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας της Επιτροπής, ώστε να λάβουν γνώση της πανδημίας και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Είδαμε τι μέτρα πρόληψης μπορεί να ληφθούν, τι ε, φαρμακευτικά μέτρα και ο οργανισμός για τον έλεγχο των ε, νόσων μπόρεσε να δώσει μια αξιολόγηση του κινδύνου και μια μελέτη για το ε, όλο θέμα. Η Επιτροπή για την Ασφάλεια της Υγείας μπόρεσε να εκδώσει σοβαρές, μια σειρά δηλώσεων για μεταξιδοτικές οδηγίες ε, με συγκεκριμένες, συγκεκριμένα μέτρα για να αναφέρω μόνο κάποια παραδείγματα. Τώρα, τι τελευταίε ημέρε υπάρχουν πολλά επικριτικά σχόλια για το πώ διαχειρίστηκαν την πανδημία οι διάφορε κυβερνήσει. Και υπάρχουν και διάφορε σφαλμένε αντιλήψει εδώ. Αντιθέτω με ό,τι δηλώθηκε στα μέσα μαζική ενημέρωση, δεν άλλαξε τον ορισμό τη πανδημία ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία ένα μήνα πριν την εκδήλωση τη πανδημία. Ορίζεται ω μια παγκόσμιων διαστάσεων ασθένεια η πανδημία στον ΠΟΕ και αυτό είναι κάτι που δεν έχει αλλάξει. Ο Δόκτωρ Τσάμπερ βέβαια έκανε σχόλια που μπορεί να αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχει αλλαγή στον ορισμό του ΠΟΕ, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Επίσης έγινε ιδιαίτερα επικριτικά σχόλια για την δαπάνη κονδυλίων σε σχέση με την αγορά εμβολίων. Πολλά κράτη-μέλη δαπάνησαν ε, σημαντικά για την αγορά εμβολίων, αλλά αυτό ήταν δικαιο, θέμα δική του αρμοδιότητα. Το πόσα και σε τι ποσότητα και σε, τι ποσά θα προμηθευτούν εμβόλια. Αυτό ήταν ένα διακανονισμό που η Επιτροπή απλώ παρακολούθησε, αλλά καθορίστηκε μεταξύ των κρατών μελών και των φορέων και των παρασκευαστών των εμβολίων. Δεν έχει λοιπόν συγκεκριμένου αριθμού για τι αγορέ από την πλευρά των κρατών μελών η Επιτροπή στα χέρια τη και αν του προσεχεί μήνε τα κάτι μέλη θέλουν να του διαβιβάσουν, εμεί θα του καλωσορίσουμε. Πάντω ήταν πολύ δύσκολο το εγχείρημα των κρατών μελών όταν έπρεπε να αποφασίσουν πόσε δόσει εμβολίων θα αγοράσουν. Μη γνωρίζοντα την τελική φύση τη πανδημία και τι τελικέ τη διαστάσει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αβεβαιότητα, τα κάτι μελη ακολούθησαν την αρχή τη προφύλαξη. Προετοιμάστηκαν για το χειρότερο ελπίζοντας να μην συμβεί. Είναι άδικο τώρα να θέτουμε να αμφιβόλω την σοφία αυτών των αποφάσεων. Τη στιγμή που τα κάτι μέλη έλαβαν αυτέ τι αποφάσει, η πρώτη του μέρη να ήταν να σκεφτούν τι πρέπει να γίνει για να προστατεύσουν του πολίτε του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά μια ενδεχόμενη και επικίνδυνη πανδημία. Πριν από λίγου μήνε μόλι, η Επιτροπή ενεργοποίησε πολλές πρωτοβουλίες για να βοηθήσει τα κάτι μελη στην όλη διαδικασία. Είχαμε με έναν διαγωνισμό πολύ γρήγορα και δημιουργήσαμε και τον εικονικό ιστότοπο για την ενημέρωση σχετικά με τα εμβόλια, ώστε να διευκολύνουμε τα κάτι μελη Πολλά κάτι επίσης συνεισέφεραν σοβαρά στην... στο σχετικό ιστότοπο του ΠΟΗ <clears throat> με διάφορα δεδομένα. Να τονίσω ότι η πανδημία δεν έχει ξεπεραστεί. Στην Δυτική Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική ο ιός ακόμη ταξιδεύει. Το ίδιο και στην Ασία και την Αφρική. Ο ιός αυτός μεταφιέζεται γενετικός και μεταβάλλεται διαρκώς. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τη δυνατότητα ο ιό αυτό, ο επένδυνο για την πανδημία, να αλλάξει σε χειρότερη μορφή. Ή, αν όλα πάνε καλά, σε μια καλύτερη. Εάν όμω πάρει χειρότερη μορφή, θα κατηγορηθούν οι κυβερνήσει γιατί δεν είχαν προμηθευτεί περισσότερα εμβόλια. Η Επιτροπή αυτή τη στιγμή κοιτάζει τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από την πανδημία ως τώρα. Τον Ιούλιο θα διοργανώσει με την Βελική Προεδρία, την Μελλοντική Προεδρία, μια συνδιάσκεψη για να ανταλλάξουμε πληροφορίες <clears throat> σε σχέση με τα εμβόλια, να συζητηθούν διάφορα ζητήματα σε σχέση με τη διαχείριση, τη κυβέρνηση, τους διαγωνισμούς, την ενημέρωση και τις διεθνείς μας σχέσεις σε τέτοια ζητήματα. Ελπίζουμε να μάθουμε περισσότερα και να βελτιωθούμε για το μέλλον. Σε σχέση με την πολιτική αυτή και τις στατικές εμβολιασμού, η Επιτροπή έχει καταστήσει ανέκαθεν σαφές ότι μια στρατηγική εμβολιασμού πρέπει να βασίζεται και στην ε, ενίοτε διαθεσιμότητα. Ο σχεδιασμό όμω τη συγκεκριμένη στρατηγική εμβολιασμού κατά του συγκεκριμένου ιού ήταν μια ευθύνη και αρμοδιότητα των κρατών μελών βάσει των δικών του πόρων. Ο ΠΟΗ και η Επιτροπή συνεχίζουν να τονίζουν ότι ο εμβολιασμό είναι ο καλύτερο τρόπο αναχέτηση τη. Αναχαιτισμό τη πανδημία. Πολλοί ε, πολίτε ακόμη κινδυνεύουν και μπορεί να ε, υποστούν σοβαρέ επιπλοκέ ή παρενέργειε από τον ιό αυτό. Ήταν τα πράγματα πολύ πιο επικίνδυνα για τι εγγύου γυναίκε και τα παιδιά. Και ξέρουμε ότι η πανδημία χτύπησε ηλικιακέ ομάδε και ομάδε του πληθυσμού που δεν φαίνονται να ήταν εκτεθειμένε ω τότε στην κλασική γρήπη. Οπότε αυτό δείχνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τη νόσου, τη ασθένεια. Η Επιτροπή τονίζει επίση ότι τα εμβόλια κατά τη πανδημία που αδειοδοτήθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όσο δυνατόν συντομότερο, έχουν άριστα πιστοποιητικά ασφάλεια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα έχουν εμβολιαστεί περίπου από 39 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 7,7% του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπεριλαμβανομένων λοιπόν 35 εκατομμύρια ανθρώπων που εμβολιάστηκαν με κεντρικό συγκεκριμένα εμβόλια από το κεντρικό κράτος συμπεριλαμβανομένων 60.000 εγγύων γυναικών και νομίζουμε ότι οι απώλειες από αυτό το σύστημα φάνηκαν ένα μελιτές. Έχω λοιπόν πλήρη εμπιστοσύνη στο σύστημα ασφάλειας ε, και στον, ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ο οποίος παρακολουθεί τόσο τα ζητήματα φαρμακοπαγρύπνησης όσο και πανδημιών. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το εμβόλιο αυτό συνεχίζει να είναι χρήσιμο κατά την καταπολέμηση του κινδύνου της πανδημίας. Το σύντομο χρονικό διάστημα που είχαμε στη διάθεσή μας έδειξε να λειτουργεί αποτελεσματικά ως προς το σύστημα που έχουμε δημιουργήσει. Μπορέσαμε εύκολα να διδοτήσουμε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο για να αντιμετωπίσουμε μια κρίσιμη κατάσταση. Κάτι τέτοιο να κάνουν και οι περισσότερε χώρε παγκοσμίω που είναι εταίροι μα. Από το 2005 η Επιτροπή λοιπόν έχει εκδώσει μια σχετική οδηγία η οποία αναθεωρείται αυτή τη στιγμή και θα προσπαθήσουμε σε μια νέα εκδοχή τη μέχρι το τέλο του χρόνου να συμπεριλάβουμε νέε προσεγγίσει βάσει των ε, διδαγμάτων που αντλήσαμε από την πανδημία H1N1. Η αποτίμηση που αυτή τη στιγμή διενεργούμε και η συνολική μελέτη που χρηματοδοτείται από τον ΠΟΗ θα μας επιτρέψει να είμαστε προετοιμασμένοι για μελλοντικά φαινόμενα αυτού του τύπου, γιατί σίγουρα θα α, ε, μας τύχουν και τέτοια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Ομολογώ ότι οι απαντήσεις σας καθόλου δεν με ικανοποίησαν. Κατά πρώτον, το πρωί άκουσα προσεκτικά τον εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος ε, παρέμβει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και παραδέχτηκε ότι υπήρχε ορισμό, αλλαγή του ορισμού της πανδημίας το 2009, πριν την ε, διακήρυξη του Ιουνίου 2009 ότι προέκυψε πανδημία. Για ξαναδείτε αυτή την ακρόαση την πρωινή, εδώ μιλάμε για τον ακραγωνιαίο λίθο του συστήματος, διότι η πανδημία κηρύχθηκε από τη στιγμή που είχαν δύο βασικά κριτήρια να συμπληρώνονται. Πρώτα απ' όλα η σοβαρότητα της ασθένειας και έπειτα η έκταση, οι διαστάσεις, δηλαδή η διασυνοριακός της χαρακτήρας. Ο κύριος Φούντα είπε ότι ότι η σοβαρότητα της ασθένειας δεν είναι πλέον το, ένα απαραίτητο κριτήριο, όσο η πρώτη εμφάνιση της, του ιού. Το κατά πόσο ο ιός ήταν νέος ή όχι είναι κάτι που το συζητάμε ακόμα, αλλά οι διαστάσεις του ήταν μεγάλες. Οπότε ήταν πιθανό να προκαλέσει ζημιές περισσότερες από ό,τι μπορούσε κανείς να υπολογίσει. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Διότι αν τώρα πανδημία είναι κάτι που το ορίζουμε βάσει ενός γεωγραφικού κριτηρίου και τις ενδεχόμενες απειλές, για θανάτους, τα πάντα επιτρέπονται. Τα εργαστήρια είναι έτοιμα να μας πουλήσουν μια πανοπλία εμβολίων. Άρα, οι βουλευτές το πρωί να σα πω ότι από πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν δίστασαν να θέσουν ε, επικριτικότατα ερωτήματα. Ποιο συμφώνησε να γίνει αλλαγή του ορισμού τη πανδημία. Αυτή ήταν η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερον, λέτε ότι εφαρμόσαμε την αρχή της προφύλαξης Ωραιότατα. εμείς είμαστε ιδεαλιστέ και περασπιζόμαστε ιδεολογικά κριτήρια. Θέλω αυτή η αρχή να μπει μέχρι και στο Γαλλικό Σύνταγμα. Αλλά τι θα πείτε για αυτή την προφύλαξη τον Απρίλιο του 2009 όταν προέκυψε το πρώτο κρούσμα του ιού. Εντάξει, η αρχή υπάρχει, προβλέπουμε ένα πρόγραμμα διαχείριση και ούτω καθεξή. Όμω αυτό που σα ε, καταλογίζω σε επίπεδο επιτροπή δεν είναι αυτό δεν είναι η εφαρμογή αυτή τη αρχή. Είναι ότι δεν παρακολουθήσατε τι εξελίξει βάσει δεδομένων. Δεδομένων που έρχονται από όλε τι χώρε του κόσμου, ιδίω από το νότιο ημισφαίριο. Διότι εκεί ο ιό είχε ήδη περάσει. Είχαμε τα αποτελέσματα τη Αργεντινή, είχαμε τα αποτελέσματα τη Αυστραλία. Και ακόμη και στι Ηνωμένε Πολιτείε, η Υπουργό Υγεία τη 5 Μαου δήλωνε ότι είναι ένα ιό που λίγο βλάπτει και δεν προκαλεί τόσου θανάτου όσο η εποχιακή γρήπη. Η επίκρισή μου λοιπόν και το ερώτημα που σας θέτω σε εσά στην Επιτροπή είναι γιατί, γιατί δεν ξανά εξετάσατε την στρατηγική σας. Να πείτε στο σύνολο των κρατών μελών, γιατί εσείς στην τελική, στην στο τέλος του λογαριασμού συντονίζετε τα κράτη-μέλη, να πείτε μην κινδυνολογείτε, μην βιάζεστε, μην παθαίνετε πανικό. Εάν θέλουμε να εμβολιάσουμε, θα εμβολιάσουμε τι πιο απειλούμενε ομάδε του πληθυσμού. Αλλά μην παθαίνουμε πανικό. Πρόκειται για έναν ιό επικίνδυνο μεν, αλλά που, δεν, που είναι καλοήθη. Οπότε μόνο 5% του πληθυσμού είχε ήδη μολυνθεί από τον ιό. Να λοιπόν το ερώτημά μου. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να σας υποβάλουν τα δεδομένα που μπορεί να έχουν στη διάθεσή τους, ώστε εσείς μετά να μετατρέψετε τη στατική σας αναλόγως. Να μπορείτε να πείτε αν χρειαστεί, δεν υπάρχει κατεπήγον χαρακτήρας, δεν υπάρχει ανάγκη, δεν το κάνατε. Σας ρωτώ λοιπόν, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων που πρέπει να ελέγχει και να αδειοδοτεί τα εμβόλια τι ρόλο παίζει. Όταν λέτε ότι είναι πολύ ασφαλή τα εμβόλια, τι ξέρετε, πώς μπορείτε να το λέτε. Ακόμη και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων λέει ότι ήταν εμβόλια πάρα πολύ ταχείας δράσης και που γρήγορα διοδοτήθηκαν. Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόληψη για τα Φάρμακα λέει ότι το, πρώτη φορά εμβόλια τόσο γρήγορα διατέθηκαν στην αγορά. Και αν δεν εγώ τι παρενέργειε δεν τι παρακολουθώ, παρακολουθώ τη, τα δεδομένα που εκδίδει ο Γαλλικός Οργανισμός Φαρμάκων, δείτε τι απολογισμό έχουμε. 2,2 δις ευρώ, δις ευρώ μας κόστησε αυτή η πανδημία, ενώ διαθέτουμε 750 εκατομμύρια σε μια πενταετία για το πρόγραμμα κατά του καρκίνου και έχουμε 3.000 ε, διαφορετικές παρενέργειες και πολλούς νεκρούς, λόγω των εμβολίων μάλιστα. Και έπειτα τι διαπιστώνω, η Πολωνία είπε λόγω χάρη δεν κάνουμε εμβόλια. Δεν θα κάνουμε εμβολιασμό. Δεν είναι ιός ε, επικίνδυνος. Καμία παρενέργεια εκεί. Άρα, πραγματικά φτάνω να αναρωτιέμαι. Είσαστε επαρκώς ενήμεροι, έχετε επαρκή γνώση, έχετε κριτική θεώρηση του θέματος ή μου λέτε η Επιτροπή είναι μία βάση ουσιαστικά είναι υποχείριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και να σας διηγηθώ και ένα έκδοτο από το 86 στην ε, Σαρντοβίλ υπήρχε μια πάλι ρήπανση της ε, περιοχής. Η Ευρώπη είχε αποφασίσει να με το Τσερνομπίλ μάλλον υπήρχε η μόλυνση από τη ραδιενέργεια και θυμάμαι τα έξοδα που είχαν γίνει τώρα βρισκόμουν στο εργαστήριο ένα μήνα μετά είχε προβλέψει προδιαγραφές και πρότυπα για τα τρόφιμα η Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε κάνει κατάσχεση τροφίμων. Είχε υπολογίσει το κάσιο αναλύτρο η Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε ορίσει τα όρια σε διαφορετικά επίπεδα από ό,τι που είχε θέσει τα όρια στο 2000 Μπεκερέλ. Και τώρα έχουμε μάθει για το Τσερνομπίλ ότι από τα 20 ε, μπεκρέλ και πάνω υπάρχει κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Τότε καλά είχαμε κάνει λοιπόν. Αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν αλλάξει με την πανδημία της γρήπης. Φαίνεται ότι η Ευρώπη έγινε μια Ευρώπη που γίνεται ουραγός, ακολουθεί τις επιταγές άλλων και να απευθυνθώ και στους συναδέλφους βουλευτές. Αν τους αφήσουμε να δρουν έτσι ανενόχλητοι, αύριο θα προκύψει πάλι κάτι ανάλογο. Νέος ιός, ε, πανικός, πρόγραμμα δράσης. Τα εργαστήρια θα είναι έτοιμα να πουλήσουν εμβόλια. Εγώ θα σας έλεγα να οργανώσουμε μια επιτροπή έρευνας, διότι αν δεν το κάνουμε αυτό ήδη από τώρα για τη διαχείριση αυτής της πανδημίας, σας διαβεβαιώ ότι αύριο θα έχουμε ένα παρόμοιο πρόβλημα και θα χάσουμε όλοι μας την αξιοπιστία ενώπιον των πολιτών της Ευρώπης οι οποίοι θα πούν ο ΠΟΗ, με τον οποίο θα υπάρχουν σίγουρα διαφορές με τα φαρμακευτικά εργοστήρια. Να σας πω ότι ο υπεύθυνος του ΠΟΗ σήμερα δεν έδωσε τους αριθμούς των ειδικών του, διότι θέλει, λέει, να διασφαλίσει το προσωπικό απόρριτο των υπαλλήλων του. Πολύ αρνητικός ήταν ο αντίκτυπος αυτού του σχολείου. Τέλος πάντων, είτε διασφαλίζουμε την αξιοπιστία των δικών μας θεσμικών οργάνων, είτε Μα σα το λέω, δεν επιτίθεμαι στην ε, Επιτροπή. Δεν είναι αυτό ο στόχο. Θέλω να βελτιωθεί η λειτουργία τη Επιτροπή, να βελτιωθεί η λειτουργία των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Διότι αν αύριο αντιμετωπίσουμε την ίδια κατάσταση, πρέπει να ξέρουμε τι θα απαντήσουμε. Πρέπει να μπορούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, έχουμε κάνει ό,τι χειρότερο για την κοινή γνώμη. Πριν σα δώσω το λόγο, κυρία Παρβάνοβα, Ξέρω ότι δεν παρεμβαίνει ο Πρόεδρος άμεσα στις συζητήσει, θέλω όμως να δώσω την, και τη δική μου θέση. Εγώ συμφωνώ απολύτως ε, με την αίτηση κοινοβουλευτική εξέτασης της Μισελ Χιβαζή. Προσωπική μου θέση είναι αυτή και νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Πιστεύω ότι είναι θεμελιώδου σημασία έναντι των Ευρωπαίων συμπολιτών μα να ασκήσουμε ε, αυτό το δικαίωμα υπέρ τη διαφάνεια. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, είδαμε και στι τελευταίε εκλογέ μπορούν να λειτουργήσουν μόνο αν έχουμε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μα. Όταν βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο οι συμπολίτε μα αντιστάθηκαν στον εμβολιασμό, που δεν ήταν ε, υποχρεωτικό βλέπουμε ότι είναι αντίσταση αλλά παράλληλα και αμφισβήτηση της πληροφόρησης που τους δόθηκε. Αν τα αφήσουμε τα πράγματα έτσι και αν αφήσουμε να θεωρούν ότι η Ευρώπη, όπως είπε η Μισελ Χιβαζή, ήταν ουραγός ή ακόμη χειρότερα ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν, ελήφθησαν επί τη βάση πληροφοριών που δεν ήταν απόλυτα αντικειμενικές, είναι σαφές ότι την ημέρα που θα έχουμε δυστυχώς ε, ε, ένα σοβαρό υγειονομικό πρόβλημα στην Ευρώπη, δεν θα μπορούμε να το διαχειριστούμε γιατί κανείς δεν θα εμπιστεύεται το λόγο των πολιτικών. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε αυτό το οποίο θέλει η δημοκρατία, δηλαδή τη διαφάνεια, αλλά παράλληλα και την ικανότητα των θεσμικών μας οργάνων να μπορούν να παρέμβουν, αν μέσα στα επόμενα χρόνια όντως υπάρξει μια σοβαρή επιδημία, πρέπει οπωσδήποτε να ρίξουμε φως στον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαχείριση αυτής της υπόθεσης. Και δεν λέω να βρούμε από δύο πομπέους τράγους και υπευθύνου, αλλά να κατανοήσουμε και να διορθώσουμε τα εσφαλμένα για να μπορέσουμε να έχουμε την εμπιστοσύνη του κοινού. Αυτά ήθελα να πω και δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Παρβανόβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν ένα διαδικαστικό θέμα πριν ε, μιλήσω για αυτό που ήθελα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και έχουμε μόνο έξι ευρωβουλευτέ, λιγότερου δηλαδή εκπροσώπου του Κοινοβουλίου από ότι εκπροσώπου τη Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να φροντίσει η Γραμματεία την επόμενη φορά να περιβρίσκονται περισσότεροι ευρωβουλευτέ στην αίθουσα. Όταν λαμβάνουμε αποφάσει για τόσο σοβαρά θέματα, για μια ειδική εξεταστική επιτροπή, θα πρέπει να καταλήξουμε στη συμφωνία, θα ψηφιστεί και στην Ολομέλεια. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να δείξουμε μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Λοιπόν, περνώ τώρα στην παρατήρησή μου. Εδώ δεν είμαστε ποινικό δικαστήριο και δεν ψάχνουμε να βρούμε κάποια θύματα, όμως είμαστε ερετοί. Όλοι μας περνάμε από δύσκολη κρίση κάθε πέντε χρόνια ε, στις εκλογές, ενώ η Επιτροπή και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν κατεβαίνουν σε εκλογές. Ούτε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νόσων ε, ε, υπόκειται σε εκλογές. Μπορεί να πάρουν σύνταξη στη θέση την οποία έχουν. Ενώ εμείς κάθε πέντε χρόνια περνάμε εξετάσεις μπροστά στους πολίτες μας. Και πρέπει να απαντάμε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα. Ερωτήματα στα οποία ζητάμε τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ε, επαρκή απάντηση. Πρόκειται και για τη διαφάνεια, πρόκειται και για θέματα λογοδοσίας και πιστεύω ότι είναι και θέμα υπευθυνότητα. Όταν ξεκίνησε αυτός ο πανικός, έγινε μια μεγάλη ακρόαση στην Ολομέλεια και καλέσαμε την Επίτροπο, την κυρία Βασιλείου τότε, που ήρθε και μας έδωσε όλα τα δεδομένα και συμφωνήσαμε ότι θα υποστηρίξουμε το σχέδιο της Επιτροπής και θα δώσουμε συστάσεις στα κράτη-μέλη για το πώς να προετοιμαστούν. Τώρα βλέπουμε ότι τα δεδομένα δεν υποστηρίζουν αυτό το οποίο δημοσιεύθηκε προς το κοινό και όλα αυτά τα μηνύματα, τα προειδοποιητικά, δεν υποστηρίχθηκαν από τεκμηρίωση, δεν τεκμηριώθηκαν και δεν είναι πρώτη φορά, είναι, έχει ξανασυμβεί. Εδώ έχουμε σημαντικά αριθμητικά στοιχεία, αλλά αν τα συγκρίνετε με τον αριθμό των κρουσμάτων της εποχιακής γρήπης θα δείτε ότι είναι τεράστιος ο αριθμός των θυμάτων της εποχιακής γρήπης. Την πρώτη φορά που είχαμε τέτοιο πρόβλημα ήταν με την γρήπη των πτηνών. Πάλι προειδοποιήσεις από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, πανδημία κλπ. κλπ. Συζητούσαμε για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε και τελικά είχαμε 270 κρούσματα με γρήπη των πτηνών σε ολόκληρο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη. Ε, είναι γελίο και αν γίνει και τρίτη φορά, νομίζω ότι θα μας βάλει σε ομοιρία μιας επικίνδυνης πρακτικής. Δηλαδή υποκείμεθα σε πιέσεις ε, από λόμπι ή από ανθρώπους που είναι να υποφελούνται από αυτό. Και αν θέσουμε το ερώτημα ποιος εποφελείται, νομίζω ότι είναι προφανές και από τα στοιχεία που έδωσε η Μισελ Ριβαζία, αν συγκρίνουμε την υπόθεση της Πολωνία, στη Γαλλία και σε άλλα κράτη-μέλη, δεν υπάρχει σημαντική προστιθέμενη αξία αυτής της δράσης που κόστησε τόσα χρήματα. Και η αποδοτικότητα, η σχέση κόστος-οφελίας, θα πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνεται υπόψη, ιδιαίτερα όταν λαμβάνουμε αποφάσεις υποπίεση. Αυτή η απόφαση και η απόφαση για την γρήπη των πτηνών ελήφθησαν υπό σοβαρή πίεση από τον κλάδο, από κάποιους ε, ιατρικούς κύκλους και από τα μέσα ενημέρωσης. Ισχυρή πίεση από τα μέσα ενημέρωσης. Υπήρχε, υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν υπήρχε κανένας λόγος να υπάρχει πανικός. Όμως ε, τα μέσα ενημέρωσης ε, πίεσαν τόσο πολύ που παρουσιάστηκε το θέμα ως πολύ πιο σοβαρό από ό,τι ήταν. Απαιτούσαν από την κυβέρνηση και από τα Υπουργεία Υγείας να δώσουν τόσα χρήματα. Και αν πάρετε αυτό το παράδειγμα της Γαλλίας για τη θέση προτεραιοτήτων, μας δείχνει ότι όταν ο Σαρκοζή ανακοινώνει το επταετές πρόγραμμα για τον καρκίνο με 750.000 ευρώ σε σύγκριση με 2,2 δισεκατομμύρια είναι, είναι, είναι γελίο. Πόσες ζωές θα σώσουμε με τόσα χρήματα. Η κοινή γνώμη ζητάει τη σωστή ισορροπία. επί δύο θητείες του Κοινοβουλίου και τώρα είναι η τρίτη θητεία του Κοινοβουλίου αγωνίζονται τα άτομα που πάσχουν από διάφορους ιούς να βρουν κάποια, κάποιο φορέα να ακούσει τα αιτήματά τους. Και τα, τα, ε, οι ασθενείς από καρκίνο επίσης ε, απαιτούν μεγαλύτερη φροντίδα. Νομίζω λοιπόν ότι αξίζει τον κόπο να δοθεί απάντηση στα ερωτήματά μας και θα συνεχίσουμε μέχρι ότου υιοθετηθεί μια συνεπής θέση. Και δεν θέλουμε να έχουμε κάποια θύματα αυτών των εξεταστικών μας κινήσεων, αλλά θέλουμε οι άνθρωποι που λαμβάνουν αποφάσεις να γνωρίζουν ότι κοστίζουν οι αποφάσεις τους και γι' αυτό θα πρέπει το κόστος και ωφέλη να λαμβάνονται υπόψη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Παρβανόβα κυρία Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ. Αντίθετα με αυτά τα οποία είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, νομίζω ότι είχαμε μόνο τα 1040 θύματα, ακριβώς διότι ελήφθησαν τα μέτρα. νομίζω ότι θα μας κατηγορούσαν πολύ περισσότερο και εμάς και την Επιτροπή αν δεν είχαμε λάβει αυτά τα μέτρα. Εγώ προχώρησα σε εμβολιασμό και των δύο παιδιών μου ακριβώς γιατί θεωρώ ότι έπρεπε, θεωρούσα ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό τον κίνδυνο. Συμφωνώ με την Υπουργό, την Προεδρεύουσα του Συμβουλίου σε αυτά που ανέφερε για την πανδημία. Πιστεύω ότι ακόμη δεν έχει παρέλθει η περίοδος της πανδημίας. Είναι πολύ νωρίς για να ζητήσουμε μια εξεταστική επιτροπή αφού ακόμη δεν έχει εξελιχθεί, δεν έχει φτάσει στο τέλος της η πανδημία. Πιστεύω ότι αυτή τη, στιγμή, αυτή τη χρονική στιγμή δεν υπάρχει κανένας λόγος να ζητήσουμε να συνταχθεί μια εξεταστική επιτροπή. Θέλει κανείς άλλο το λόγο? αλλά όχι να ξαναδώσω λόγο στον κύριο ρή. Ευχαριστώ πολύ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όλες αυτές οι ερωτήσεις απασχολούν και μας. Δεν είμαστε υπάλληλοι που κάθονται και πληρώνονται για να μην κάνουν τίποτα και να μην δρούν. Εργάζομαι κι εγώ και ελπίζω ότι σκέφτομαι κιόλας. η πολύ καλή ερώτηση, ε, μάλλον ε, να το θέσω όλος, θα προσπαθήσω να εστιάσω σε κάποια ε, στοιχεία. Η κυρία Ριβαζή αναφέρθηκε στις αλλαγές τους ορισμούς. Ο ορισμός της πανδημίας είναι τμήμα ενός τελείως μεγαλύτερου ε, πακέτου διεθνών κανονισμών. Συζητήθηκε το 1999 με την πρώτη οθέτηση το 2005 και το 2009. Δεν βλέπουμε όμως κάποια σχέση μεταξύ της αλλαγής του ορισμού και της λογικής της ανακοίνωσης της πανδημίας. Η σοβαρότητα ενός περιστατικού δεν συζητήθηκε ποτέ ως τμήμα της όλης διαδικασίας ε, και δεν ξέρω κατά πόσον εμείς θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και επίσης θα ήθελα να δούμε και τον ορισμό της πανδημίας ως τμήμα της διαδικασίας. Διότι υπάρχει τέταρτο, πέμπτο και έκτο επίπεδο πανδημίας. Ε, ε, το είπε και ο Πόη, το είπε και ο καθηγητής Τσάτ. Αλλά υπάρχει και αυτό που είπε η κυρία Κάντεμπαχ όλες οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συμφώνησαν ε, σε ένα σχέδιο ετοιμότητας και ε, όταν ξεκίνησε η πανδημία κάθε κυβέρνηση συνέχισε με το εθνικό της σχέδιο και την εκτέλεση ουσιαστικά όλων όσων είχαν συμφωνηθεί νωρίτερα. Έχουμε λοιπόν ορισμό πανδημίας, έναρξη του 5ου και 6ου επίπεδου και εθνική δράση. Και αυτό φυσικά είναι το πιο σημαντικό σημείο που πρέπει να συζητήσουμε στη διάρκεια της περίοδου αξιολόγησης. Ε, χθες ο κύριος Τσάτ μας είπε ότι θα ξεκινήσει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση. το κατά πόσον παρακολουθήσαμε τα όσα συνέβαιναν στο νότιο ημισφαίριο. Φυσικά, παρακολουθούμε στενά τα πράγματα αυτά, διότι έχουμε εμπειρογνώμονες που εργάζονται για μας, ε, για τον ε, Ευρωπαϊκό Φορέα ε, και όλοι θέλουμε να ξέρουμε περισσότερα πράγματα για τον ιό. Αλλά όταν μελετά κάποιος την κατάσταση, η εικόνα δεν είναι πολύ σαφής. Ε, το Μεξικό, για παράδειγμα, στο Νότιο ημισφαίριο είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ε, στο Μεξικό έχουμε τρεις, ε, ε, τρία κύματα ε, επιδημίας του ιού. Ε, στην Ευρώπη έχουμε μόνο ένα κύμα. Αυτή είναι η κατάσταση τουλάχιστον. Αλλά στο Μεξικό βρισκόμαστε ήδη στο τρίτο κύμα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε γιατί υπάρχει σχέση με τη θερμοκρασία και τον ιό αν είναι η χαμηλή θερμοκρασία αυτή που επιδεινώνει την κατάσταση. Αυτά όλα είναι ασαφή. Και φυσικά η εικόνα που έχουμε από το νότιο ημισφαίριο δεν ήταν μεν ισχνή, αλλά δεν απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες, Αμερικανοί, Ιάπωνες εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε με όλα όσα έχουν ε, συμφωνηθεί στο σχέδιο τιμότητας. Όσον αφορά τώρα στη στρατηγική εμβολιασμών, αυτό και πάλι ήταν απόφαση εμπειρογνωμόνων από τα κράτη-μέλη, από τον από το Κέντρο Προέλευση Νόσων. Ε, όλα αυτά ε, γίνανε με κάποια επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη. Δεν τα αποφάσισε η Κομισιόν από μόνη τη. Ε, όλα αυτά είναι στη φάση της ανάπτυξης. είναι και θέμα στρατηγικής. Σε πολλές χώρες αποφασίστηκε να εμβολιαστούν μόνο κάποιες συγκεκριμένε ευάλωτε ομάδες, όχι όλοι. Άλλε χώρε προσέφεραν εμβόλια για όσους πολίτες ήθελαν να εμβολιαστούν. η σχέση τώρα μεταξύ της ε, στρατηγικής που συμφωνήθηκε για τον εμβολιασμό και η εκτέλεση. Και αυτή είναι μια σημαντική ε, παρατήρηση. Ε, υπάρχει χώρα της Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία μπορεί να πάτε και να δείτε ότι έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό εμβολιασμού. Η εκστρατεία πήγε καλιά και έγινε πολύ και την αποδέχτηκε ο πληθυσμός. Ε, ξέρουμε για παράδειγμα ότι και στον Καναδά είχαμε πολύ υψηλό ε, επίπεδο εμβολιασμών ε, του πληθυσμού, αλλά σε άλλες χώρες δεν ήταν και τόσο ευπρόσδεκτοι από τους πολίτες. Διότι διαπιστώνουμε ότι προσφέρθηκαν μεν τα εμβόλια, δεν υπήρχαν επικρίσεις, δεν μας δίνεται εμβόλια, υπήρχε θέμα προσωπικής επιλογής. Θέλω να εμβολιαστώ ή δεν θέλω να εμβολιαστώ. Και φυσικά καμία κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένη να κάνει υποχρεωτικό εμβολιασμό. Γι' αυτό ακριβώς και δεν έχουμε υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ούτε καν συζητήθηκε κάτι τέτοιο. Τώρα, το θέμα της αξιολόγησης των εμβολίων. Θα μπορούσα να σας ζητήσω, σας παρακαλώ, ζητώ συγγνώμη κύριε Διευθυντά, αλλά ε, οι διερμηνείς θα πρέπει να σταματήσουν στις 6 και μετά. Είναι δυνατόν λοιπόν να ολοκληρώσετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ολοκληρώσω. Στο θέμα τη διαφάνεια. Στι αρχέ είμαστε πολύ ανοιχτοί για ενημέρωση. Υπήρχε πάντα εκπρόσωπο κάθε μέρα, ο οποίο ήταν διατεθειμένο να απαντήσει σε ερωτήσεις. Είμαστε διατεθειμένοι να ενημερώσουμε το κοινό, τις κυβερνήσει, Ήμασταν σε στενέ επαφέ με διάφορου φορεί ε, από διεθνεί οργανώσει και θέλαμε να συλλέξουμε και γνώσεις αλλά και να ενημερωνόμαστε όσο το δυνατόν περισσότεροι. Στο τέλος όμως αξιολογήσαμε το κόστος και το όφελος. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ε, θέμα συζήτησης, διότι ελπίζω ότι όταν θα ολοκληρωθεί το θέμα της πανδημίας να δούμε και τι ωφέλη αποκομίσαμε από αυτό. Δεν είναι σαφές ε, αυτό που είπε και η κυρία Κάντεμπαχ τι ακριβώς άλλαξε την όλη εικόνα. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί και καταφέραμε να διατηρήσουμε την πανδημία υπό έλεγχο. Να υπενθυμίσω ότι δύο χώρες, ε, το Μεξικό και η Ουκρανία, είχαν πολύ μεγάλα προβλήματα και αυτή την εικόνα την κρατήσαμε κι εμείς. Ε, το Μεξικό γιατί ήταν η πρώτη χώρα και η Ουκρανία για πολλούς άλλους λόγους. Αλλά η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική ε, ανάλογα με την ανταπόκριση της κάθε ε, χώρας. Στην αρχή βέβαια για το Μεξικό τα πράγματα ήταν δύσκολα γιατί όπως σας είπα ήταν η πρώτη χώρα και ε, Εκεί ήταν λίγο δύσκολο να αντιδράσουν, τους έπιασε εξαπίνης ο ιός, αλλά για την Ουκρανία ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Η... Το γεγονός ότι διαβιβάζονταν λοιπόν οι πληροφορίες ήταν πάρα πολύ καλό και οι επόμενοι μήνες θα είναι ένα πολύ καλό διάστημα για αξιολόγηση, για περισυλλογή και φυσικά είμαστε διατεθειμένοι να μοιραστούμε όλες αυτές τις πληροφορίες με το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε αύριο στις 9 για τις ψηφοφορίες. Καλό βράδυ.